Uh, good morning everyone. First point, adoption of the... Καλημέρα σας. Πρώτο σημείο, η εγκρίση της διάταξης. Εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσει, εγκρίνεται. Ευχαριστώ. Σήμερα το πρωί έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Αρίας Καλνίτε. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ σήμερα. θα συζητήσουμε την πρόταση για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και τα πρότυπα για τα οχήματα, τα αυτοκίνητα και τα φορτηγάκια κατά την έναρξη των εργασιών μας. Είμαι βέβαιη ότι οι συγκητές μας θα εργαστούν σκληρά για να βεβαιωθούν ότι αυτό το νέο νομοθέτημα θα μας βοηθήσει να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει των συμφωνιών τη Συμφωνία των Παρισίων και για να μειώσουμε τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα στα ελαφρά εμπορικά οχήματα και στα τηλεοπτά. Ευχαριστούμε κύριε Πετροπέ, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, ευχαριστώ για την πρόσκληση να σα παρουσιάσω σήμερα τι νομοθετικέ προτάσει Τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής για τα πρότυπα εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα για το διάστημα μετά το 2020, για τα ελαφρά εμπορικά και τα γιοταχή. Σα ευχαριστώ για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε και για την πολύ καλή δουλειά που έγινε στις τρεις κύριες προτάσεις για να πετύχουμε στόχου, ε, στόχους μείωσης του 40% στο 2030. Στο σύστημα ανταλλαγής εκπομπών ε, το διοξιδίου του άνθρακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και στο Λουλουσιεφ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Χερμπράντι, την κυρία Γκίρλινγκ και τους σκιώδεις εισηγητές καθώς και όλους όσοι συμμετείχαν στην προσπάθεια αυτή διότι η ολοκλήρωση των εργασιών μας θα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την υλοποίηση των ε, δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη Συμφωνία των Παρισίων. Ταυτόχρονα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Τέλη για τον διορισμό της ως για την πρόταση των εκπομπών διοξείδου του άνθρακα από τα αυτοκίνητα και τα φορτηγάκια και θέλω να συνεργαστώ μαζί της και με τους κοιόδης εισηγητές και όλη την Επιτροπή σας. Για να είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρξει ταχεία πρόοδος σε αυτό το θέμα που είναι υψηλής πολιτικής σημασίας. Με περίπου ένα τέταρτο των συνολικών εκπομπών της Ευρωπαϊκή Ένωση να προέρχονται από τις συγκοινωνίες. Ο τομέας αυτός έχει έναν ζωτικό ρόλο διαδραματίσει στη μετάβαση σε μια ε, οικονομία απαλλαγμένη από τον άνθρακα. Ε, η Ευρώπη έχει μειώσει τις εκπομπές της κατά 23% από το 1990. Οι οδικές μεταφορές όμως έχουν διωγγωθεί κατά 20%. Σήμερα οι εκπομπές από τις μεταφορές είναι περίπου το 22% του συνολικού ποσοστού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι μεταφορέ συνεχίζουν να εντείνονται και να αυξάνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η νομοθετική πρόταση τη Ευρωπαϊκή Ένωση που προβλέπει νέα πρότυπα για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγάκια μετά το 2020 είναι θεμελιώδε ε, σημασία. Σήμερα θέλω να επικεντρωθώ στα τρία βασικά στοιχεία αυτής της νομοθετικής πρότασης. Πρώτον, το επίπεδο φιλοδοξιών και το χρονοδιάγραμμα για τα πρότυπα του διοξιδίου του άνθρακα και δεύτερον τα κίνητρα και τους μηχανισμούς για τις μηδενικές εκπομπές και τα οχήματα χαμηλών εκπομπών. Και τέλος τη νέα βελτιωμένη διακυβέρνηση και τους κανόνες επιβολής. Ε, να ξεκινήσω με τους στόχους ε, διοξιδίου του άνθρακα και το χρονοδιάγραμμα. Η πρόταση θέτει ρεαλιστικούς στόχους για τα πρότυπα για τα αυτοκίνητα και φορτηγάκια και για το 2025 και για το 2030 και βασίζεται σε μια συνολική ανάλυση μαζί με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και των εκπροσώπων του κλάδου των παραγωγών ο στόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το μέσο όρο εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα θα πρέπει να είναι 30% χαμηλότερο στο 2030 σε σύγκριση με το 2021. Η πρόταση επίση περιλαμβάνει και έναν ενδιάμεσο στόχο μείωσης 15% για το 2025 και για τα αυτοκίνητα και για τα φορτηγάκια. Αυτό θα μας ε, εξασφαλίσει ότι οι επενδύσεις θα ξεκινήσουν δυναμικά ήδη τώρα. Ενώ ο στόχο για το 2030 μα δίνει έναν μακροπρόθεσμο ορίζοντα, τον οποίο θα πρέπει να σεβαστούμε σε σχέση με αυτέ τι ε, ε, φιλοδοξίες. Τα πρότυπα δίνουν μια κατεύθυνση για τις συγκοινωνίες και για να μπορέσουμε να επιδιώξουμε του συμφωνημένο μας στόχου βάσει της συμφωνίας των Παρισίων. Η πρόταση αυτή μαζί με τα νέα πρότυπα για τα φορτηγά, τα βαρέα οχήματα που θα υποβάλουμε στις 2 Μαΐου θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη να επιτύχουν τους δεσμευτικούς τους στόχους βάσει του κανονισμού για την κατανομή των προσπαθειών καταναλωτές στην Ευρώπη θα υποφεληθούν από το μειωμένο κόστος κατανάλωσης καυσίμων και από καλύτερη ποιότητα στην ατμόσφαιρα, στον ατμοσφαιρικό αέρα. Επίσης θα υπάρχει γενικό θετικό αντίκτυπος για την απασχόληση επειδή επιτρέπει μια ε, ομαλή μετάβαση σε χαμηλές εκπομπές και μηδενικές εκπομπές καθώς και τα οχήματα που θα τις προκαλούν. Για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτύχει τους κλιματικούς και ενεργειακούς της στόχους για το 2030 βάσει των δοσμεύσεων της Συμφωνίας των Παρισίων και για τους μακροπρόθεσμους στόχους απαλλαγής από τον άνθρακα τα οχήματα με μηδενικέ και χαμηλέ εκπομπέ θα κερδίσουν ένα σημαντικό μερίδιο τη αγορά. Γι' αυτό το λόγο, μαζί με του στόχου για το διοξίδιο του άνθρακα, η νομοθετική πρόταση περιλαμβάνει ένα νέο καινοτόμο σύστημα παροχή κινήτρων, ώστε οι αυτοκινητοπαραγωγοί να έχουν περισσότερα καθαρά ε, οχήματα και φορτηγά στην αγορά, στη διάθεση τη αγορά, στην ερχόμενη δεκαετία. Η πρόταση θέτει δείκτε ε, συγκριτική αξιολόγηση για το πόσα καθαρά οχήματα κάθε αυτοκινητοπαραγωγό θα πρέπει να έχει παράγει στο το 2025 και 2030. Όταν οι παραγωγοί παράγουν περισσότερα καθαρά οχήματα πάνω από του δείκτε, τότε θα πάρουν περισσότερες πιστώσεις ε, για την επίτευξη των στόχων διοξιδίου του άνθρακα. Ο μηχανισμός κινήτρων είναι ε, ουδέτερος ως προς την τεχνολογία. Καλύπτει όχι μόνο τα οχήματα με μηδενικές, αλλά και των χαμηλών εκπομπών οχήματα και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ομαλή μετάβαση προς την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών. Κάνει διάκριση μεταξύ των οχημάτων βάσει των επιδόσεών του ως προς το διοξίδιο του άνθρακα και ε, τα οχήματα με μηδενικές εκπομπές που καταμετρώνται ε, πλήρω, σε ένα πλήρε ποσοστό, ενώ αυτά των χαμηλών εκπομπών μόνο εν μέρη. Το σύστημα αυτό θα επιτρέψει στου αυτοκινητοπαραγωγού να περάσουν σε καινοτόμε λύσει και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά του. Η πρόκληση τη βιώσιμη κινητικότητα είναι πολύ σημαντική στη ζήτηση για καθαρά προϊόντα, τεχνολογίε και επιχειρηματικά μοντέλα. Και είναι μια τεράστια επιχειρηματική ευκαιρία για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και την, τον μηχανικό τη κλάδο. Η επιτυχία των ε, οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών δεν θα βοηθήσει ε, δεν θα σχετιστεί μόνο με τους στόχους που θα θέσουμε, αλλά και με το κατά πόσον διατίθεται υποδομή για την επαναφόρτιση. Και επίσης, κατά πόσον οι μπαταρίες και η γρήγορη φόρτιση θα είναι σε ανταγωνιστικές τιμέ στην αγορά. Έτσι, για να έχουμε την ε, ανανέωση των υποδομών, το πακέτο της καθαρής κινητικότητας περιλαμβάνει και ένα πρόγραμμα δράσης με ε, μέτρα ε, επενδύσεων για την ανά την Ευρώπη ε, ανάπτυξη υποδομών για εναλλακτικά καύσιμα ε, με 800 εκατομμύρια αξία. Αυτό είναι απαραίτητο για να αποφύγουμε το δίλημα της κόταση του αυγού που εμποδίζει την αγορά καθαρών οχημάτων από τους καταναλωτές και να είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρχουν σταθμοί επαναφόρτησης και για τα καύσιμα Βεβαίω, είναι σημαντικό να υπάρχουν ανταγωνιστικέ τιμέ και για τι μπαταρίε. Γι' αυτό θα πρέπει να πάρουμε πίσω την παραγωγή μπαταριών στην Ευρώπη και να είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον αγώνα για τι μπαταρίε επόμενη γενιά. Είναι σημαντικό για την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση η Ευρώπη να έχει τη δυνατότητα να παράγει ε, φτηνότερε και καλύτερε μπαταρίε ω καύσιμα για τα οχήματα του μέλλοντο. Έτσι λοιπόν η πρωτοβουλία για τι μπαταρίε που έχει ε, ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα συμβάλλει σε μια ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε τα οχήματα και άλλε λύσει τη κινητικότητα για το αύριο και τα και διάφοροι παράμετροι τη να αναπτυχθούν και να παράγονται στην Ευρώπη. Το τρίτο στοιχείο τη πρόταση είναι η καλύτερη επιβολή των κανόνων. Θέλουμε να μην υπάρχουν πλέον κενά και να βεβαιωθούμε ότι οι καταναλωτέ ε, εποφελούνται όπω ε, του υποσχεθήκαμε. Το όλο σύστημα θα βασίζεται στο νέο κύκλο για τα τεστ των αυτοκινήτων το εναρμονισμένη, την εναρμονισμένη διαδικασία τεστ για τα ελαφρά οχήματα που ελπίζουμε ότι θα έχει πιο ακριβείς και ρεαλιστικές μετρήσεις. Ωστόσο η νομοθεσία θα είναι αποτελεσματική μόνο να βεβαιωθεί ότι οι τιμές των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα από τα τεστ είναι ορθές και αντιπροσωπευτικές των ε, εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες. Γι' αυτό θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα από συστήματα κατανάλωσης των καυσίμων που θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά σε όλα τα νέα οχήματα. Έτσι θα βεβαιωθούμε ότι η μείωση των εκπομπών είναι κάτι που αποτελεί πραγματικότητα και όχι μόνο μία θεωρητική ιδέα. Η πρόταση επίσης προβλέπει τεστ συμβατότητας για να βεβαιωθούμε ότι τα οχήματα που παράγονται είναι τόσο καθαρά όσο αυτά που δοκιμάστηκαν. Οι αποκλήσει θα ανοιχνεύονται και αυτό θα λαμβάνεται υπόψη κατά την επαλήθευση των ε, στόχων συμβατότητα των αυτοκινητοπαραγωγών. Αυτά τα νέα μέτρα συμβαδίζουν πλήρω με τι συστάσει του Μηχανισμού Επιστημονικών Συμβουλών καθώ και με όσα μα σύστησε το Ευρωκοινοβούλιο μετά τι ε, έρευνε τη Επιτροπή ΕΜΗΣ. Εν είδη συμπεράσματο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει μια φιλόδοξη και ρεαλιστική πρόταση που πιστεύουμε ότι ε, επιτυγχάνει το σωστό σημείο ισορροπία μεταξύ περιβαλλοντικών ε, ε, στόχων και στόχων για του καταναλωτέ και την απασχόληση. Ανεπομονούμε για να συνεχίσουμε την εξαιρετική μα συνεργασία φέτο για την πρόταση αυτή και να έχουμε μια ταχεία έγκρισή τη πριν το τέλο αυτή τη θητεία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Θα έχουμε δύο γύρους ερωταπαντήσεων. Στον πρώτο γύρο θα ακούσουμε τους συντονιστές ή τους εκπροσώπους τους. Θα έχει δύο λεπτά ο καθένας. Ο κύριος Μπέλετ καταρχάς. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και καλή σας ημέρα. Επίτροπε, θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ. Αναφερθήκατε στην καλύτερη εφαρμογή και επ' αυτού έχω μια ερώτηση πράγματι τα οχήματα που κινούνται στους δρόμους θα πρέπει να έχουν τις ίδιες επιδόσεις στο δρόμο με αυτές που έχουν στο εργαστήριο. Αυτό είναι προφανές. Άρα, όπως και μας είπατε, θα εξαρτηθεί η επιτυχία των μέτρων από το πόσο σωστές είναι αυτές οι δοκιμές και είπατε ότι οι κατασκευαστές θα πρέπει να βάλουν στα νέα οχήματα αυτές τις συσκευές μέτρησης καυσίμων έχουμε και την οδηγία για την έγκριση των οχημάτων που συνιστά πρόοδο και θα μετρήσει πολύ και αυτή για την επιτυχία και της εποπτείας από πλευράς κομισιών που πρέπει να αναλάβει την εποπτεία για το πώς εφαρμόζονται οι εθνικοί κανονισμοί. Μπορείτε να μας εγγυηθείτε ότι οι απάτες του παρελθόντος δεν θα επαναληφθούν και ότι όλα τα κενά και παραθυράκια πράγματι θα κλείσουν. Δεύτερο ερώτημα, αν με επιτρέπετε, κυρία Πρόεδρε. Το δεύτερο ερώτημα, κύριε Επίτροπε, αφορά αυτές τις αποκαλύψεις ε, των τελευταίων ημερών στον τύπο. Δεν έχουν άμεση σχέση με τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, αλλά έμεσα συνδέονται τερά, ε, μάλλον ε, πολύ φοβερές αποκαλύψεις ε, για πειράματα σε πυθίκους, ίσως και σε ανθρώπους από ό,τι φαίνεται, για να μετρηθούν τα αποτελέσματα που έχουν και ο αντίκτυπος που έχουν εκπομπές στην υγεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισήμως αντέδρασε, το γνωρίζω αυτό. Θα ήθελα, αφού είστε εδώ όμως, να ακούσω και την προσωπική σας άποψη τα ναι, νέα αυτά είναι τρομακτικά και φρικτά. Μπορεί να λάβει μέτρα η Κομισιόν για να αντιμετωπιστούν αυτού του είδους οι πρακτικές και να μην ξαναγίνουν κάτι αντίστοιχο στο μέλλον. Ευχαριστώ κύριε Μπέλετ, ο κύριος Ντάνς. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και τον Επίτροπο. Εκ μέρους της κυρίας ε, Μίρια Μντάλη μιλώ εγώ. Όπως γνωρίζετε, είναι εισηγήτρια για τη νέα νομοθεσία σε σχέση με τι εκπομπέ δεξιοτάρια τα οχήματα. Από τότε που ε, δημοσιεύθηκε η μέτρο για την κινητικότητα, φαντάζομαι ότι έχετε διαβάσει τα σχόλια ε, και δει τα σχόλια τη ομάδα μα ότι είμαστε υπέρ οποιοδήποτε μέτρου θα μειώσει τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Βέβαια, θα πρέπει να έχετε επίση υπόψη ότι είμαστε και κάπω ε, επικριτικοί απέναντι στο πεδίο εφαρμογή και το εύρο και το φιλοδοξία του πακέτου. Πολλά περισσότερα πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη για να φτάσουν του στόχου του 2030 δυνάμει του κανονισμού για την επιμερισμό των προσπαθειών και οι οδικέ μεταφορέ συνεισφέρουν τα μάλιστα στι εκπομπέ. από τομεί που δεν καλύπτονται από το ETS για την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών. Ε, υπάρχουν ανησυχίε ότι αν οι εκπομπέ των οδικών μεταφορών συνεχίσουν να αυξάνονται, θα αντισταθμίσουν πλήρως τις μειώσεις άλλων ε, τομέων. Και φυσικά οι τομείς αυτοί κάναν πάρα πολύ σοβαρές προσπάθειες. Δεν κάνει αυτά που θα έπρεπε ο τομέας των οδικών μεταφορών για να επιφέρει τι απαιτούμενε μεταφορές ε, και να πληρωθούν οι στόχοι που έχουμε θέσει. Για να έχουμε λοιπόν αυτές τις εκπομπές θα πρέπει να είναι πολύ καλύτερες οι επιδόσεις των οχημάτων και χρειάζονται νέοι στόχοι. Όσο το δυνατόν πιο γρήγορα πρέπει να εφαρμοστούν. Πρέπει τα ηλεκτρικά οχήματα να είναι ένα σημαντικό κομμάτι του στόχου οχημάτων μέχρι το 2030. Και επίσης για να κλείσουμε τα κενά θα μπορούσαν οι αδίστακτοι κατασκευαστές να εκμεταλλευτούν και τα παραθυράκια. Ξέρετε ότι είμαστε υπέραυστηρών στόχων. Το Κοινοβούλιο και η ομάδα εργασία του Κοινοβουλίου έχει εργαστεί επ' αυτού του θέματο. Αλλά το ερώτημά μου, κύριε Επιτροπή, είναι πώ η Κομισιόν θα εξασφαλίσει ότι η διαδικασία λήψη αποφάσεων κατά τι διοργανικέ διαπραγματεύσει θα διευκολυνθεί και τι σχέδια έχετε επ' αυτού. Γιατί αυτή η νομοθεσία πρέπει να ολοκληρωθεί και να περατωθεί επιτυχώ ω το δυνατόν πιο γρήγορα για να αρχίσει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2020. Εσεί έχετε ένα χρονοδιάγραμμα, δηλαδή πότε θέλετε να έχουν ολοκληρωθεί όλε οι διαπραγματεύσει. Πρόεδρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Ντέμες Μάκερ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Επίτροπο για τις εξήγησεις που μας έδωσε. Φαντάζομαι γνωρίζετε πως ε, ήμουν αντιπρόεδρος ε, της Εξεταστικής Επιτροπής και αν θέλουμε να δείξουμε ότι υπάρχει σαφής δέσμευση υπέρ της δημόσιας υγείας, ε, και βέβαια της οικονομίας, είναι σημαντικό να υιοθετήσουμε πιο αυστηρά πρότυπα που όμως θα μπορούν και να εφαρμοστούν και να επιβληθούν αποτελεσματικά. Και όπως είπατε και εσείς δεν θα πρέπει να μείνει στα χαρτιά η πρόταση αλλά να μεταφραστεί στην πράξη πρόταση αυτή μας δίνει πραγματικά τη δυνατότητα να βελτιώσουμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα πιο αυστηρά πρότυπα είναι κάτι αναγκαίο και φέρνουν και ωφέλη, προωθούν ε, τις επενδύσεις στην καινοτομία και ανοίγουν το δρόμο σε ένα τεχνολογικός ουδέτερο πρασίνισμα του στόλου οχημάτων. Επίσης ε, θα βοηθήσουν στην εξοικονόμηση καυσίμου, άρα θα ε, είναι και καλά νέα για το πορτοφόλι των καταναλωτών. Πιο αυστηροί κανόνε είναι κάτι που πρέπει να το στηρίζουν και τα ίδια τα κρατημέλη. Γιατί έτσι θα μπορούν ε, να υιοθετήσουν και αντικειμενικού ε, κλιματικού στόχου με την βοήθεια και τη σύγχρονη τεχνολογία. Νομίζω ότι η δέσμη μέτρων αυτή παρέχει σχετικέ ευκαιρίε. Σε ό,τι αφορά τα επιβατικά οχήματα και τα φορτηγάκια λέμε ότι η μείωση των διεξιδίων του του άνθρακα μέχρι το 2030 δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί. Το κόστος για τους καταναλωτές είναι πιο χαμηλό από ό,τι πιστεύω σε σχέση με το 2020 αυτούς τους στόχους. Τα είχε πει στην Επιτροπή ΕΜΗ τον Ιούλιο του 2016 ένας τέος και συγκεκριμένα είχε πει ότι οι κατασκευαστές οχημάτων έχουν συμφέρον να υπολογίσουν το κόστος συμμόρφωσης πριν την έγκριση του κανονισμού, γιατί το υψηλό κόστος θα μπορούσε να κάνει τους ρυθμιστές να αποδυναμώσουν ή να εγκαταλείψουν τον προτινόμενο κανονισμό. Και έπειτα θα μπουν σε μια κούρσα μείωση του κόστου συμμόρφωσης στο ελάχιστο. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να απαντήσετε, να αντιδράσετε σε αυτή τη δήλωση. Εγώ προσωπικά Θέλω να συνεισφέρω με θετικό τρόπο ώστε να έχουμε μια δέσμη κανόνων αποτελεσματική για να μειωθούν ε, οι εκπομπές εξιδίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, κύριε Κανιέτη που βρίσκεστε εδώ μαζί μας. Θα ήθελα να ζητήσω ε, συγγνώμη που η φωνή μου είναι λίγο βραχνή Χαιρόμαστε φυσικά που βλέπουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χαιρόμαστε που βλέπουμε το δευτερεύοντα στόχο. Αλλά δεν μας ικανοποιεί η φιλοδοξία της. Ε, στη Φιλανδία ε, διεξάγουμε μια ε, μελέτη ιδιωτική αφορά τα κίνητα οχήματα δεύτερης γενιάς για περικοπή των ε, εκπομπών κατά 90% ε, ε, σχεδόν. Όταν εσείς λέτε περικοπή κατά 30% θεωρούμε ότι η φιλοδοξία σας υπολείπεται. Εμείς προσεγγίζουμε το πρόβλημα τα διαφορετικά. Οπότε θα ήθελα να μου πείτε τι άλλε οδοί υπάρχουν, διότι υπάρχει τρόπος ε, συνδυασμού των διαφόρων τεχνολογιών ώστε να μπει κανεί πιο γρήγορα στο μέλλον με καθαρότερα οχήματα. Θα ήθελα επίσης να μας πείτε κατά την άποψή σας πώς θα συμβάλλει αυτή η πρόταση στο συνολικό στόχο ε, των ε, συμφωνιών του Παρισιού. Όπως είπαν και οι άλλοι ομιλητές, ε, μας ανησυχεί το ότι το ότι δεν είναι αυτή που θα έπρεπε. Θα θέλαμε λοιπόν να μας το αναλύσετε λίγο παραπάνω. Επειδή τελειώνει ο χρόνος μου και εξασθενίζει και η φωνή μου, θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τόρβαλτς. κύριε Κονέτσινα. αξιότιμη επίτροπε, αντίθετα από τους συναδέλφους, εγώ καταλαβαίνω τις προσπάθειές σας να μην θέσετε υπερβολικά φιλόδοξους στόχους. Γιατί τελικά ε, οι πολύ φιλόδοξοι στόχοι δεν ε, οδήγησαν σε κάτι θετικό, αλλά στο σκάνδαλο του Dieselgate. Θα πρέπει λοιπόν να, να είμαστε λογικοί και να εξασφαλίσουμε ότι οι στόχοι θα μπορούν να, να εφαρμοστούν στην πράξη συνολικά και όχι να παραμείνουν στο χαρτί. Εδώ ε, πρέπει να ξέρουμε ότι η νομοθεσία αυτή πρέπει να είναι λογική. Δεν το βλέπω όμως στην προκειμενομική πράξη ό,τι αφορά τις διαφορές των πραγματικών εκπομπών και των εκπομπών στο εργαστήριο. Όλο και μεγαλώνει το χάσμα, το, η ψαλίδα και επίσης ε, για την ε, ε, δαπάνη η οποία αυξάνεται 400 ευρώ το χρόνο για τα καύσιμα τα, οποία πρέπει, τα χρήματα αυτά πρέπει να δίνουν οι καταναλωτές. Σίγουρα είναι σημαντικό να μειωθούν αυτές οι διαφορές. Αλλά δεν νομίζω ότι θα έχουμε επιτυχία και θα είναι όλο και πιο υψηλές οι τιμές σε σχέση με στο δρόμο από ό,τι στις, ε, στα εργαστήρια. Δεν θα το πετύχουμε αυτό το στόχο μέχρι το 2030. Θα είναι πολύ ψηλές εκπομπές στο δρόμο, κατά την άποψή μου. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν αυτήν την ε, διαφορά μεταξύ του τι ισχύει στο χαρτί και του τι ισχύει στην πραγματικότητα. Αυτή τη διαφορά πρέπει να την ε, διατηρήσουμε στο δυνατόν πιο μικρή σε ό,τι δεν αφορά ε, τις ε, δοκιμές σε πραγματικέ συνθήκες οδήγηση, Πρέπει να τι βελτιώσουμε και οι κατασκευαστές ε, οχημάτων θα πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσει για τιμή των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Κύριε Επίτροπε, η Κομισιόν είχε προετοιμάσει αυτό τον κανονισμό ε, για τα αυτοκίνητα και τα ελαφριά φορτηγά και στη σχετική μελέτη. Κατάληξαμε στο συμπέρασμα ότι για να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης κατά 60% των εκπομπών μέχρι το 2050 η απόδοση των οχημάτων και των ελαφρών φορτηγών πρέπει να βελτιώνεται κατά 6% ετησίω. Επίσης, τόνισαν ότι έχοντα το νου μα τη συμμόρφωση με το Παρίσι θα πρέπει να υπάρξουν ακόμα καλύτερες βελτιώσει. Ταυτόχρονα εκτιμάται ότι οι μεγαλύτερες εξοικονομήσεις κόστους τόσο για την κοινωνία στο σύνολό τη, όσο και για του τελικού χρήστε, επιτέχθηκαν με τους αυστηρότερους στόχους το Διεθνές ε, Συμβουλίο Καθαρής Μεταφοράς, ε, Καθαρών Μεταφορών καταλήξει το συμπέρασμα μάλιστα ότι τα ωφέλη για την κοινωνία και για τους καταναλωτές θα είναι καλύτερα με μείωση του διοξιδίου του άνθρακα κατά 70% μέχρι το 2030. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε για ποιο λόγο η Κομισιόν αποφάσισε μείωση του στόχο μείωσης του διοξιδίου του άνθρακα που δεν συνάδει ούτε με τους στόχους ε, της Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2050 ούτε με τις ε, ε, δεσμεύσεις ε, της Συμφωνίας του Παρισιού και που δεν οδηγεί ταυτόχρονα στα μεγαλύτερα δυνατά ωφέλη για την κοινωνία. Και η δεύτερη μου ερώτηση σχετίζεται με αυτό. Οι υποθέσει κόστου τη Κομισιόν όσον αφορά τη βελτίωση της απόδοση των καυσίμων συμβατικών κινητήρων είναι πάνω από το ICCT. και δεν συνάδουν και με τα πορίσματα της ε, συμβουλευτική εταιρεία που ανέλησε τα δεδομένα για την Κομισιόν. Και μου φαίνεται, όπως ε, ρώτησε και η συναδελφός, ότι όχι μόνο η αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι ειλικρινής ε, στην ανάλυση των δυνατοτήτων μείωσης κόστους που θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει ο κανονισμός. Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς έχετε καταλήξει σε τέτοιες ε, ε, υποθέσεις κόστους στην πρόταση αυτή. Ευχαριστώ κυρία Εύη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα Επίτροπε. Δυστυχώς ε, για άλλη μια φορά διακρίνω μια κομισιόν που δείχνει, επιδεικνύει δύναμη με τους αδύναμους και αδυναμία με τους ισχυρούς. Ε, να εξηγήσω, αυτές τις μέρες ε, είδαμε τις ακροάσεις πολλών υπουργών περιβάλλοντος από όλη την Ευρώπη που διαρκώς ε, παραβιάζουν τους κανόνες ποιότητας του αέρα και δικαίως η Κομισιόν παρεμβαίνει και καταλήγει στην τελική φάση όπου θα εκδώσει ένα πρόστιμο μέσω του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και που φαίνεται ότι θα είναι πολύ ψηλό ε, στην Ιταλία, μάλιστα, τα πρόωρα θύματα λόγω της ατμοσφαιρικής ρήπανσης ε, είναι, ε, έχουν τον υψηλότερο αριθμό στην Ευρώπη. Ναι, αυτές οι παραβιάσεις πράγματι θα πρέπει να τιμωρηθούν και θα όμως κοστίσουν πολλά στα κράτη-μέλη και στις τσέπες των πολιτών. Μου φαίνεται ωστόσο από την άλλη πλευρά ότι οι προτάσεις που κάνει η Κομισιόν, αυτή είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος, οι προτάσει που εφαρμόζει για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα τη ποιότητα του αέρα, ειδικότερα στον τομέα των μεταφορών, δυστυχώ είναι πολύ αδύναμε. Εγώ συμμερίζομαι τι επικρίσει ορισμένων συναδέλφων. Πράγματι, δεν είναι αρκετά φιλόδοξη αυτή η πρόταση. Το στόχο του 30% ακόμη και βάσει άλλων επιστημονικών δεδομένων είναι πολύ χαμηλός και διαφωνώ. Δεν μου αρέσει αυτός ο μηχανισμός ε, που προτείνεται που δεν θα λειτουργήσει αυτός ο μηχανισμός ε, ε, τιμωρίας ε, των κατασκευαστών που δεν θα επιτύχουν τους στόχους. Πιστεύω δεν θα φέρει αποτελέσματα. Για άλλη μια φορά μου φαίνεται ότι φιλοδοξία της Κομισιόν δεν είναι επαρκής. Δεν μπορεί λοιπόν να έρχεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον κακό συνέχεια προσπαθώντας να αυξήσει ε, το φιλοδοξίο και τελικά να προσκρούσει παρά το των κρατών μέλων στο Συμβούλιο, όπου φυσικά τα κράτη-μέλη θα κάνουν οτιδήποτε για να μειώσουν τη φιλοδοξία αυτή. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, εδώ ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος. Ε, έχετε το λόγο κύριε Πίτροπε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συντονιστές οι οποίοι παρενέβησαν στη συζήτηση αυτή. Και αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι αυτό το ζήτημα. Χρειάστηκε πολύ χρόνο ε, για να εκπονήσουμε στην Κομισιόν ε, το έγγραφο αυτό. Από εξωτερικού συμβούλου πήραμε πολλέ πληροφορίε, είχαμε εκατοντάδε συναντήσει με ΜΚΟ και άλλου ενδιαφερομένου φορεί πριν καταλήξουμε στην πρότασή μα. Κάποιοι λέτε ότι δεν είναι αρκετά φιλόδοξοι. Να σα πω όμω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει τη όλα τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα για να εκπώνησε αυτή την πρόταση. Έχουμε μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία σε ό,τι αφορά ε, τις θέσεις εργασίας που προσφέρει. Είναι θεμελιώδης δε για κάποια κράτη-μέλη. Πρέπει να βελτιώσουμε την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέριου τους πολίτες. Πρέπει να έχουμε οχήματα χαμηλών εκπομπών, πρέπει να έχουμε την κατάλληλη υποδομή για τις μπαταρίες και όλα αυτά πρέπει να τα κάνουν ταυτόχρονα και έχουμε και τους στόχους της συμφωνία του Παρισιού που πρέπει να πληρώσουμε. Σας το λέω τη εξ αρχής, γιατί κάποιοι ασκήσατε μια κριτική για το στόχο του 30% που είπατε ότι δεν είναι αρκετά φιλόδοξο σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία του Παρισιού. Έχω να σας πω το εξή. Όταν έκανε τις προτάσεις για το Λουλουσιεύ, για τον πεσμό των προσπαθειών, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλα αυτά τα έκανε στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει, ακριβώς στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Παρισίων. Σε τις ε, εθνικές μας ε, συνεισφορές και από όλους τους κλάδους, από όλους τους τομείς. προτάσεις μας νομίζω ότι επιτυγχάνουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ τριών βασικών στόχων Πρέπει να τους δούμε ταυτόχρονα. Ε, αντίκτυπο στο περιβάλλον, υπηρεσίε προ καταναλωτέ και αντίκτυπο στην απασχόληση. Το 30% τη μείωση για το περιβάλλον πιστεύω ότι θα βοηθήσει να μειωθούν οι στόχοι ε, για το 2030 στον τομέα των κτηρίων της Γεωργίας και σε αυτούς τους τομείς που δεν καλύπτουν από το ETS. Είπατε οι μεταφορές πρέπει να κάνουν πολλά. Ναι, πρέπει. Αλλά και τα κτίρια πρέπει να κάνουν πολλά στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης. Είμαστε αφιλόδοξοι με το στόχο 3% για την ενεργειακή απόδοση και άλλοι τομεί λοιπόν θα είναι φιλόδοξοι στον κανονισμό για τον πρισμό των προσπαθειών. Δεν λέμε ακριβώ τι πρέπει να κάνει το κράτο μέλο ε, για τον κάθε τομέα, γιατί εξαρτάται αυτό από τι ιδιαιτερότητε του κάθε κράτου μέλου. Οι μεταφορέ δεν είναι ακριβώ ε, το ίδιο στην Αυστρία ε, με τη Μάλτα και την Κύπρο, γιατί υπάρχουν ιδιαιτερότητε. Βέβαια, το αναλυτικό έργο. όταν κατατέθηκε η πρόταση για τον επιμερισμό προσπαθειών, δείχνει ε, ότι θέλουμε να έχουμε μία μείωση κατά 25% των εκπομπών για τις οδικές μεταφορές. Και αν δείτε τα αποτελέσματα των ε, στόχων μας ε, και των μέτρων, θα έχουμε μείωση 22% για το 2030. 25% έλεγε το αναλυτικό έργο για μείωση των εκπομπών. Για όλο τον τομέα των μεταφορών και όχι μόνο για τα ελαφρά εμπορικά οχήματα και τα αυτοκίνητα. Η πρόταση, μάλλον το αναλυτικό μέσα μας λέει ότι θα φτάσουν στο 22% και το 3% που απομένει από τα πρότυπα για τα φορτικά που θα προτείνουμε το Μάιο θα επιτευχθεί. Πρέπει να τα δούμε από κοινού όλα αυτά. Και έτσι θα φτάσουμε στο επίπεδο που θέλαμε. Σύμφωνα με τη στρατηγική μας. Αν δείτε αυτή τη μείωση του 40%. Φυσικά να δείτε μόνο την ε, περιβαλλοντική πτυχή, ε, όσο μειώνεις ε, τόσο έχεις πρόβλημα με τη στρατηγική για την απλή από άνθρακα. Τι γίνεται όμως ε, με τις πολιτικές για την απασχόληση. Μείον 30, μείον 40. Ποια είναι η διαφορά. 3%. Γιατί μπορείς να μειώσεις όσο θέλεις. Αλλά μετά επηρεάζεις τους προμηθευτές, την αυτοκινητομηχανία, άρα και την απασχόληση. Άρα πώς μπορούμε να είμαστε αποδοτικές προς το κόστος. Ένα άλλο ερώτημα ήταν η Κομισιόν τι ρόλο έχει να διαδραματίσει στην όλη αυτή διαδικασία. Τον ίδιο ρόλο που παίζαμε μέχρι τώρα. Είμαστε οι διαμεσολαβητές μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Πιο φιλόδοξο το Κοινοβούλιο από το Συμβούλιο. Εμείς είμαστε ο έντιμος διαμεσολαβητής μεταξύ των δύο. Επίσης, αν μας λέει το Κοινοβούλιο και μας ρωτάει ποια είναι η επίπτωση του να έχουμε παραδείγματος χάρη επίπεδο μείωσης 50% τι επιπτώσει θα έχει αυτό στην απασχόληση ή για το περιβάλλον τι επιπτώσει θα έχουν αυτά τα μέτρα. Ό,τι τεχνική πληροφορία και ό,τι στοιχεία χρειαστεί και ζητήσει το Κοινοβούλιο θα του τα δώσουμε, θα τα ε, παραγάγουμε αυτά τα στοιχεία και θα βοηθήσουμε και την τους νομοθέτες να πάρουν σόφρονες αποφάσεις. Έχουμε πάρα πολλούς λομπίστες που επηρεάζουν. Μελετήσαμε όμως πάρα πολλές ε, εκθέσεις και μελέτες και ε, εκατοντάδες ε, έγγραφα. Και θέλαμε μετά να δούμε και με τους κατασκευαστές και τους προμηθευτές ποιο είναι το κόστος και τι δυνατότητες υπάρχουν. Αναλύσαμε πάνω από 80 διαφορετικές τεχνολογίες και το κόστος κάθε μιας σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των καταναλωτών. Ο στόχος το 30% θα είναι επωφελής για όλους τους καταναλωτές. Θα πρέπει να πληρώσουν πιο υψηλέ τιμέ για τα πιο αποδοτικά οχήματα καταναλωτέ. Μεν, όμω αυτό θα αντικατασταθεί από άλλε εξοικονομήσει για νέα οχήματα. 600 ευρώ για ένα όχημα που αγοράστηκε το 2025 και έως 1.500 ευρώ για ένα όχημα που αγοράζει ο καταναλωτής το 2030. Αν έχουμε τον στόχο του 40% αυτή η αντιστάθμιση πάβει να ισχύει. Και οι μελέτες αντικτύπου λένε ότι το 40% θα μειώσει τα ωφέλη για τους καταναλωτές και την κοινωνία. 300 ευρώ για ένα μέσο όχημα. Το κόστος για τους καταναλωτές θα αυξηθεί κατά 800 ευρώ ένα όχημα. θα επηρεαστεί και η απασχόληση. Έχουμε ένα πρόβλημα εδώ. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε μια ομαλή μετάβαση σε οχήματα χαμηλότερων εκπομπών. Και βέβαια πρέπει να εξασφαλίσουμε και ένα επαρκή ένα επαρκές χρονικό διάστημα για να επανεκπαιδευτούν ή να αναποκτήσουν νέες δεξιότητες οι εργαζόμενοι στον κλάδο της αυτοκινητομηχανίας. αύξηση ηλεκτρικών οχημάτων. Ναι, σίγουρα όλα αυτά είναι καλά, αλλά θα αλλάξει τελείω η αλυσίδα εφοδιασμού. 300 εξαρτήματα έχει ένα ηλεκτρικό όχημα. Αλλά ένα συμβατικό όχημα έχει 1300 εξαρτήματα. Θα επηρεαστεί λοιπόν πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό έχουμε καταθέσει αυτή την πρόταση. Για τα υβριδικά οχήματα που έχουν ρόλο στην ένταση εργασίας, γιατί έχουν κλασικοί μηχανισμοί ε, έγχυσης ε, και καύσης, καυσίν. Η μετάβαση πρέπει να γίνει προοδευτικά. Γι' αυτό δεν πάμε κατευθείαν στα μηδενικών εκπομπών οχήματα, αλλά έχουμε αυτό το ευρεδικό μοντέλο ως ε, μεταβατική λύση, που έχει και δυνατότητα φόρτισης, δηλαδή. Ακούστε τώρα κάτι άλλο. Η Τσεχία πάνω από το το 2,8, 2,1 Ρουμανία έχουν το θέμα της απασχόλησης. Δηλαδή αυτά τα ποσοστά που σας είπα είναι εργαζόμενοι στον τομέα αυτό και θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Και για την ομαλή μετάβαση πρέπει να φροντίσουμε, όπως είπα θα γίνει επίσης με τις δομές επαναφόρτησης των οχημάτων. Θυμάστε τι έγινε όταν συζητούσαμε την οδηγία για τα κτίρια. Δεν υπήρχε αρκετή φιλοδοξία για τις υποδομές τότε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θέλουμε πιο φιλόδοξους στόχους. Προετοιμάσαμε, αυτό ήταν ο στόχος μας, νομίζω μια ισορροπημένη πρόταση. για να αποφύγουμε τα λάθη του παρελθόντος. Έχουμε εισαγάγει δύο νέα στοιχεία. Γιατί είναι σαφέ τι έχει αλλάξει. Ο κύκλος ε, δοκιμών στο HLDP. Αλλά αυτό επίσης είναι εργαστηριακή δοκίμη και υπάρχει ένα κενό μεταξύ εργαστηριακής δοκιμής ε, και δοκιμής σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Να μην αυξηθεί αυτό το κενό, αυτό θέλουμε αυτή η ψαλίδα. Και έχουμε εισαγάγει δύο νέα στοιχεία για την ενίσχυση των ελέγχων. Καταρχάς ένα νέο εργαλείο παρακολούθησης ε, των ε, εκπομπών. Το WLTP θέλουμε να παραμείνει αντιπροσωπευτική δοκιμή. Αυτό το εναρμονισμένο παγκοσμίω ε, πρόγραμμα δοκιμών για ελαφρά οχήματα. Θέλουμε να έχουμε και αυτή τη χαμηλή τεχνολογίας για τη μέτρηση του καυσίμου. Θέλουμε να υπάρχει τυποποιημένη κατανάλωση καυσίμου μέσω της ειδικής σε όλα τα οχήματα για να μπορούμε να μελετάμε, να υπολογίζουμε την κατανάλωση καυσίμου και να βλέπουμε τι γίνεται. Ποιο είναι το κενό μεταξύ πραγματικότητα και του WLTP. Δεν θέλουμε να αυξηθεί, αλλά να μειωθεί, τουλάχιστον παραμείνει στάση αυτή τη διαφορά. Και ένα άλλο στοιχείο είναι πόσο αντιπροσωπευτικό είναι αυτό το σύστημα. Θα παίρνουμε στοιχεία συνεχώς και θα τα ομαδοποιούμε και θα τα δημοσιοποιούμε. Αυτό είναι το σημείο. Θα τα δημοσιοποιούμε. Άρα οι καταναλωτέ έχουν στη διάθεσή του έτσι ένα νέο εργαλείο για να καταλάβουν ποια είναι η κατανάλωση, μάλλον ποια είναι η επίδοση του καυσίμου, ώστε να έχουν να πληρώσει αυτό που πήραν. Και έχουμε και τις δοκιμές συμμόρφωσης ε, για τις εκπομπές ε, του άνθρωπου ώστε οι καταναλωτές να έχουν αυτό που πληρώνουν. Και τα οχήματα που κατασκευάζονται να είναι πραγματικά ε, όσο καθαρά φαίνεται να είναι στα εργαστήρια και στο δρόμο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην τριμερή διάλογο στήριξε σχετικές απόψεις. Είχαμε όμως μια τελική πρόταση για την έγκριση τύπου που δεν συμπεριέλαβε αυτή την διάταξη. Γι' αυτό και την ξαναεντάσσουμε σε αυτόν τον νέο κανονισμό και ελπίζουμε ότι θα μας υποστηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε τελικά να υιοθετηθεί. Υπήρχε και μια συγκεκριμένη ερώτηση για το κόστος και πώς υπολογίζεται και τι συνέβη την περασμένη φορά. Οι προβλέψεις μας για το κόστος βασίστηκαν σε 10 μελέτες, σε διεξοδική μελέτη αντικτύπου και τη διαρκή συνεργασία με το αρμόδιο κέντρο για να αξιολογήσουμε τις νέες τεχνολογίες. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι μάθαμε τι έγινε στο παρελθόν από τις διάφορες παρεκκλήσεις στο εκτιμόμενο κόστος. Τώρα αυξήσαμε το επίπεδο ακρίβειας για να μην γίνουν και άλλα λάθη. Έγινε και μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση για τα κίνητρα. Εδώ η πρόταση περιλαμβάνει έναν μηχανισμό ε, κινήτρων για τα, μηδενικά, για τα οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών. Διότι δεν θέλουμε να μείνουμε πίσω στον όλο αγώνα δρόμου για τα οχήματα αυτά. Αυτή τη στιγμή έχουμε 1% νέε πωλήσει τέτοιων οχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα ο καταναλωτή τη Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ε, διαλέξει από ένα πολύ περιορισμένο αριθμό τέτοιων οχημάτων, ενώ στην Ασία έχουν 400 επιλογές. Σήμερα λοιπόν οι επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνε στην Καλιφόρνια, την Κίνα, επειδή και έχουν ισχυρότερα κίνητρα, έχουν ποσόστοση ηλεκτρικών αυτοκινητών για το 2019-2020 στην Κίνα, με 7 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα στόχο παραγωγής μέχρι το 2025. Το ρυθμιστικό μας μήνυμα για το μέγεθο τη αγοράς που να πετύχουμε στο μέλλον θα δώσει το κατάλληλο ε, κίνητρο στους επενδυτέ και στου ε, ιδιωτικού και δημόσιου ε, παροχή για τις υποδομέ επαναφόρτηση. Ελπίζουμε ότι θα δώσει επίση το κατάλληλο μήνυμα. Κάποιοι από εσά είπαν γιατί δεν επιβάλλουμε και κάποιε κυρώσει, κάποιε ποινέ σε σχέση με το επίπεδο ηλεκτροκινητών οχημάτων και αν δεν αυτό δεν επιτευχθεί. Ένα σύστημα δηλαδή που και μπόνους να δίνουμε και να επιβαλούμε και κάποιο πρόστιμο. Ε, έχουμε χαράξει το δρόμο για ένα τέτοιο σύστημα ενδεχομένως, αλλά στην πράξη θέλουμε να έχουμε πρώτα ένα στόχο, ένα πλαίσιο. Τώρα θα μου πείτε Γιατί η Επιτροπή δεν έχει προβλέψει κάποιο τέτοιο, κάποια εντολή συγκεκριμένη. Μπορεί κανείς να προβλέψει εντολή, δηλαδή υποχρέωση που να συμπεριλαμβάνει κυρώσεις και πρόστιμα, αλλά χρειάζονται και τα εργαλεία για να υπάρξει πραγματική ε, παρουσία των ηλεκτροκινητών οχημάτων. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει εντολή, φορολογικά κινήτρα και η αναλόγη πολιτική για να υπάρξουν σταθμοί επαναφόρτηση. Όμω για να επιβληθεί μια τέτοια εντολή υποχρέωση στου αυτοκινητοπαραγωγού δεν έχουμε. Αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να δοθούν κίνητρα από το κυβερνητικό επίπεδο για να διευκολυνθεί η αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων ή οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών, και αν επίση δεν έχουμε την άμεση δυνατότητα να αναπτύξουμε υποδομές επαναφόρτησης δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια υποχρέωση εντολή. Δεν μπορούμε να την προβλέψουμε. Σίγουρα θα υπάρξουν ε, ποινέ εάν το κινητοπαραγωγή δεν ε, συμμορφωθούμε με του στόχου για το διοξείδιο του άνθρακα. Αυτού που έχουμε θέσει. Διότι εκεί οι τεχνολογίε υπάρχουν, είναι διαθέσιμε, όμως για να υπάρξει η ανάπτυξη, η διάδοση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, ικανοποιηθεί και η ζήτηση των ε, καταναλωτών αφού πρώτα σου καλλιεργηθεί, πρέπει πρώτα να υπάρξουν και δημόσιοι στόχοι. Για τα υβριδικά οχήματα, α πούμε, υπήρχε ένα σταθμό επαναφόρτηση. Και με τέτοιου είδου πρόταση, αυτό ο στόχο δεν έγινε αποδεκτό από το Κοινοβούλιο. Γι' αυτό αυτό το σύστημα με τα πριμ και τα, τις ποινές δεν έγινε αποδεκτός. Επίση, έγιναν κάποιες ερωτήσεις για τις πρόσφατες ειδήσει. Για τα τεστ περί εκπομπών σε ζώα και ανθρώπους. Όπως φαντάζεστε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πάθει σοκ με αυτέ τι ειδήσει. Όπως κάθε άλλος. Ελπίζουμε ότι οι γερμανικές αρχές ε, κάνουν έρευνα στο θέμα. Είναι αρκετά σαφές ότι οι δοκιμές ε, στα ζώα δεν θα πρέπει να υπάρχουν καν στην Ευρώπη. Εργαζόμαστε προς αυτόν τον στόχο και κοιτάζουμε να εγκρίνουμε εναλλακτικέ διαδικασίες για να συμβεί αυτό. Οι δοκιμέ στα πειράματα σε ζώα αυτή τη στιγμή υπόκειται σε τρομερά αυστηρού κανόνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρούμε ότι θα πρέπει να, μειωθούν να μειωθούν σταδιακά και να εξαλειφθούν πλήρω. Όσο για τα πειράματα σε ανθρώπου, θα πρέπει να γίνει έρευνα. Σας ευχαριστούμε για αυτό το γύρο ερωτήσεων. Θα περάσουμε στον επόμενο και θα σας παρακαλέσω τώρα να παραμείνετε στο ένα λεπτό. Πρώτος, η κυρία Γιούζο. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Οι στόχοι μου φαίνονται λογικοί, αλλά το σημαντικό είναι να επιτευχθούν. Οι εκπομπές έχουν να κάνουν με το βάρος του οχήματος, με τις νέες τεχνολογίες που θα μπουν στόχοι. Και όλο και πιο μεγάλο χήματα θέλουν οι καταναλωτές. Η μάζα ε, είναι όγκος, ένα κριτήριο για την Κομισιόν και τι άλλα κίνητρα θα μπορούσε να δώσει για να μειωθεί ε, τουλάχιστον στις πόλεις ε, το μέγεθος, η διαστάση του χήματος. Τώρα, είπατε ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά και πραγματικά. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει και αυτές οι μετρήσεις και τα μέτρα να είναι και διαφανή και να δημοσιοποιούνται σε τακτά διαστήματα τα στοιχεία αυτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά την τροποποίηση οδηγία για την επισήμανση ε, των οχημάτων, σε ό,τι αφορά τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Το αποτύπωμα άνθρακα των ε, εξαρτημάτων των οχημάτων δεν θα πρέπει να καλύπτει όλο το χρόνο ωφέλιμης ζωής, παραδείγματος χάρη, οι μπαταρίες. Για την κατασκευή τους απαιτούνται σημαντικές εκπομπές δείξετε το άνθρακα. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε. Ο κύριο Πανιού. Ναι κύριε Επιτρόπε, δύο λόγια, κάποιες ερωτήσεις και να εκφράσω την εκτίμησή μου για τις προσπάθειές σας στους τομείς ε, αρμοδιότητάς σας από το 2014. Ελπίζω ότι το χέρι σας ε, έτσι όπως είναι δεμένο δεν θα παρεμποδίσει τη δυναμικότητά σας ε, έτσι όπως την έχουμε διαπιστώσει και εδώ και εγώ ως εισηγητής για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για την COP21 και σε διάφορες περιστάσεις. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι το αριστερό σας χέρι λειτουργεί μια χαρά. Οπότε αυτό είναι καλό σημάδι, κύριε Επίτροπε. Σημαίνει ότι το νομοθετικό πακέτο για την καθαρή κινητικότητα που παρουσιάζεται φαίνεται θα φέρει καλά αποτελέσματα για το μέλλον σε ένα πλαίσιο όπου φυσικά πρέπει να νομοθετήσουμε. Αποτελεί μεγάλη ανησυχία για τους Ευρωπαίους και τις Ευρώπες ε, το όλο θέμα αυτό, όλα τα προβλήματα υγείας των συμπολιτών μας προβλήματα υγείας που οφείλονται στα οχήματα και στην κυκλοφορία, ειδικότερα στις μεγάλες πόλεις μας. Όπως βλέπουμε και εδώ στις Βρυξέλλες, για παράδειγμα. Έχω κάποιες παρατηρήσεις και κάποιες συστάσεις να σας κάνω, κύριε Επίτροπε, όσον αφορά τον κανονισμό που αφορά τους νέους κανόνες, ε, μείωση των εκπομπών, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να δείξουμε μεγαλύτερη φιλοδοξία και να ανεβάσουμε το στόχο στο 40% από το 30% μέχρι το 2030. Επίσης πιστεύω πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταματήσουν οι πωλήσει καινούριων αυτοκινήτων που εκπέμπουν αέρια θερμοκηπίου μέχρι το 2040. Να δώσουμε ισχυρά κίνητρα για την ηλεκτροκίνηση και αποτρεπτικά κίνητρα σε περίπτωση μη τήρησης των κανόνων. Να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα λοιπόν στις αυτοκινητοβιομηχανίες. Αυτά κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Παρνιό. Κύριε Μάισνερ. Um, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Κύριε Επίτροπε, πολλές ε, φορές ε, αναφέρεστε στην ηλεκτροκίνηση. Πράγματι είναι μια πολύ καλή λύση ε, εκπέμπει λιγότερα αέρια, είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον, αλλά αυτό εξαρτάται από το που έρχεται ο ηλεκτρισμός. Η παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος δεν είναι πάντα αηφόρος. Και κάτι άλλο που δεν άκουσα, ε, δεν ξέρω αν θέλετε να ακούσετε την ερώτησή μου κύριε Επίτροπε, μάλιστα, κάτι που δεν ε, είδα εδώ είναι τι άλλο γίνεται σε άλλα κράτη-μέλη για την επίτευξη των στόχων. Για παράδειγμα αναφέρατε ότι η κατάσταση διαφέρει από κράτο μέλο σε κράτος μέλο. και ειδικότερα στη Βόρεια Ευρώπη έχουμε πολύ CNG οργανικά ε, βιολογικά απόβλητα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίμων και χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα. Ε, αν έχουμε δημιουργήσει την εναλλακτική υποδαμή για καθαρότερη ενέργεια, εξετάζουμε την ηλεκτροκίνηση, το CNG, το πεπιεσμένο φυσικό αέριο και το υδρογόνο. Πρέπει να δούμε λοιπόν ε, τι δυνατότητες έχουμε παραγωγής ε, βιολογικού, βιολογικού καυσίμου. Ευχαριστώ κυρία Μάισνερ, κυρία Τόρες Μαρτίνες. Gracias. Ευχαριστώ. Γνωρίζουμε ότι μιλάμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα ρήπανσης. 400.000 άτομα χάνουν ε, τη ζωή τους ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό. Το δέσμη μέτρων ε, για την κοινικό θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε για να λυθεί αυτό το ζήτημα δημόσια υγεία, ε, αυτό το πρόβλημα τη ρήπαση στην Ισπανία. Κύριε Κανιέτα, το πρόβλημα είναι πιο σοβαρό, όπω ξέρετε, γιατί εμεί έχουμε ε, ξεπεράσει τα μέγιστα, τι μέγιστε οριακέ τιμέ και ο Υπουργό Περιβάλλοντο κατηγορούσε του Δήμου τη Μαδρίτη και τη Βαρκελόνη, επειδή μπορεί να τιμωρηθεί με πρόστιμο, επειδή δεν τηρείται οι οριακέ αυτέ τιμέ η Ισπανία. Και έβαζε ως παράδειγμα ακριβώς αυτά τα μέτρα της Δημάρχου της Μαδρίτης ε, για να καταπολεμήσει τις υψηλές εκπομπές όπως περιορισμοί, κυκλοφορία, στάθμευση, ταχύτητα των οχημάτων. Και τότε είχε δεχθεί δρυμία κριτική από τους συντρόφους ε, της, από το Λαϊκό Κόμμα για αυτά τα μέτρα. Θα ήθελα λοιπόν, ε, κύριε Κανιέτε, να σας ρωτήσω γιατί θα ήθελα να μου απαντήσετε. Πιστεύετε ότι η Μανουέλα Καρμέν δίκιο είχε και πρέπει να μειωθεί η κυκλοφορία. Γιατί εκεί εστιάζει βασικά το πρόβλημα και για τα οξύδια του αζότου και για τη ρήπανση γενικώ και την, ε, τον έφος στις μεγάλες πόλεις. Ευχαριστώ. Ο κύριο Τόμας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε λέει ο κύριος ε, Τούρμες. Ε, σας εύχομαι καλή ανάρρωση γιατί θα χρειαστεί να μαχηθείτε σε αυτόν τον αγώνα. Ο αγώνας αυτός θα έχει σκοπό να κάνει την Ευρώπη πάλι μεγάλη για τους πολίτες της, σημαντική για τους πολίτες της ε, ή να κάνει τον ντίζελ σημαντικό. Θα είναι λοιπόν μια μάχη μεταξύ του λόμπι που μάχεται για... και μας κλέβει με τον ντίζελ εδώ και μια δεκαετία και το σκάνδαλο δεν είναι κάποιοι πήθηκοι, αλλά εκατομμύρια πολίτες που εκτίθενται σε επιβλαβή αέρια σήμερα στην Ευρώπη. Αυτό είναι το σκάνδαλο. Και τι κάνει η Κομισιόν για να φύγουν από τους δρόμους αυτά τα εκατομμύρια διζελοκίνητα οχήματα από τους δρόμους και μετά υπάρχουν οι πολίτες αυτοί που πιστεύουν ότι η Ευρώπη θα πρέπει να είναι το μέρος της σύγχρονης βιομηχανίας. Το μέλλον των αυτοκινήτων θα είναι ε, η διασύνδεση και η ηλεκτροκίνηση. Αλλά το ερώτημα είναι θα παράγονται αυτά τα αυτοκίνητα στην Ευρώπη. Και ζητώ συγγνώμη, η πρόταση της Κομισιόν πολύ ωραία δεν διασφαλίζει όμως ούτε το κλίμα μας ούτε την προστασία μας από τη ρήπανση ούτε δίνει ένα μέλλον στη βιομηχανία μας. Δεν μπορούμε να καλέσουμε τους κύριους Ζάλμα και τον κύριο Βίσμαν σε αυτή την επιτροπή, κυρία Πρόεδρε, γιατί και αυτοί έχουν κάποια επιρροή ε, στην εκπόνηση των προτάσεων της Κομισιόν. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριος Γκίζη, και ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και θέλω να ευχαριστήσω και τον ε, Επίτροπο. Δεν θέλουμε να παίζουμε θέατρο εδώ, αλλά να μιλάμε αντικειμενικά για τις εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρωπου και για αυτό να και άλλα θέματα. Ε, πραγματικά ε, δεν μου άρεσε αυτή η συζήτηση μέχρι τώρα. Είπατε κάποιες προτάσεις και είπατε ότι πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές και φιλόδοξοι. Το 30% μέχρι το 2030 και 15% ε, ενδιάμεσο στόχος νομίζω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση αυτή η στόχη. Επίσης θέλουμε να τονίσουμε την ηλεκτροκίνηση. Χρειαζόμαστε καλές υποδομές ε, και για την επαναφόρτιση. δύο εκατομμύρια σταθμούς. Εγώ νομίζω ότι όταν ε, θα είναι επιδότηση μόνο 400 ευρώ αναστήλη φόρτισης νομίζω ότι τα διαθέσιμα κονδύλια δεν είναι επαρκή. Και πραγματικά όλος αυτός ο χαμός και αυτό η μοσιότητα που έχουν πάρει τα ηλεκτρικά οχήματα, μόνο εάν είναι από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το ρεύμα θα είναι ε, κάτι θετικό. Μην ακολουθούμε αυτές τις ε, αναδαφικές προτάσεις των ε, πρασίνων. Ευχαριστώ. Thank you. Mr. Terms. If Mr. Would read ο κύριος Γκύρη και να διαβάσει τις τροπολογίες μου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα δει ότι υπάρχει τροπολογία και την έχουμε ψηφίσει και αυτό ζητούμε. Όλα τα ηλεκτρικά οχήματα στην Ευρώπη να κινούνται με πράσινη ηλεκτρική ενέργεια. Μη λέτε λοιπόν λάθη και ψέματα. My name. Uh, Mr. Γκίζικη, είναι το όνομά μου, Κλόντ, όχι Γκύρε και ούτε το όνομά μου δεν ξέρεις. Λοιπόν, να στηρίσουμε τη διαδικασία. Κύριε Επίτροπε, πάντα έτσι είναι ενθουσιασμένα τα μέλη όταν έρχεστε. Ας επιστρέψουμε στους ομιλητές μας που έχουν γραφεί για σήμερα. Ο κύριος Ντάνς, ε, συγγνώμη, ε, δεν ήθελα να παρέμβω. Είναι πολύ διασκεδαστικά όλα αυτά. Δεν ξέρω αν έχουν τελειώσει. Ε, Λοιπόν, θα μιλήσω ως ευρωβουλευτές. Ε, αναφέρατε για το πόσο σημαντική είναι η αυτοκινητοβιομηχανία στα κράτη-μέλη. Ε, στο δικό μου κράτος αποφασίσαμε με το Brexit να την καταστρέψουμε. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Είναι πολύ σημαντική βιομηχανία για πολλές χώρες η αυτοκινητοβιομηχανία. Αλλά εκεί υπάρχει ο κίνδυνος να μείνουμε πίσω διότι όπως είπατε δεν υπάρχουν οι απαραίτητε υποδομές, η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές δεν έχει ακόμα επιτευχθεί, αλλά το βασικό πρόβλημα που έχουμε είναι ότι τόσο στη ΣΥΠΑ όσο και στην Κίνα υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο δυνάμεις που διασφαλίζουν την ύπαρξη των υποδομών ε, θέτουν και ανώτατα όρια και εφαρμόζουν εμπορικέ πολιτικέ ώστε να διασφαλίσουν τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα. Τι μπορεί συνεπώ να κάνει η Κομισιόν γιατί στην Ευρώπη η υποδομή ε, ελέγχεται σε εθνικό επίπεδο. Τι μπορεί να κάνει η Κομισιόν για να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη ώστε να υπάρξουν πλαίσια στο μέλλον που θα διασφαλίζουν ότι τα κράτη-μέλη έχουν τη σωστή υποδομή, διότι αν δεν το κάνουμε αυτό, θα καταστραφεί η αυτοκινητοβιομηχανία και θα βρίσκεται αλλού τελικά στο μέλλον, αντί να βρίσκεται στι χώρε μα. Και αυτό θα ήταν τραγικό. Ευχαριστώ. Κύριε Πέτερλα. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, εγώ υποστηρίζω τη στρατηγική σας, την καλωσορίζω και επίσης το ίδιο και τις φιλοδοξίες σας. Η στρατηγική που μας προτείνεται συμπεριλαμβάνει πολλές διαφορετικές στρατηγικές στην ουσία και έχει και ένα πολύ υγιές στοιχείο ευρωκεντρικού χαρακτήρα. Είναι πολύ σωστές οι φιλοδοξίες σας, ε, πολύ εύστοχες σε σχέση με τις μπαταρίες, αλλά πρέπει στην Ευρώπη να προσπαθήσουμε να παράγουμε τα καλύτερα ηλεκτροκίνητα, ηλεκτροκίνητα οχήματα στον κόσμο. Το ίδιο συμβαίνει και με τα αεροσκάφη, οπότε να φροντίσουμε και στα ηλεκτροκίνητα οχήματα να αναλάβουμε πρωταγωνιστικό ρόλο. Εγώ είμαι φιλόδοξος από τη φύση μου και πιστεύω ότι αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Το Τέσλα το ίδιο γεννήθηκε στην Ευρώπη. Ε, και επίση χαίρομαι που αναφέρατε και την ε, σχέση προ του καταναλωτέ όλων αυτών των προτάσεων. Ε, η αυτοκινητοπαραγωγή είναι πολύ καλά ε, οργανωμένη, το ίδιο και οι εργαζόμενοι, αλλά καμιά φορά οι καταναλωτέ είναι αυτοί που μένουν στην απέξω. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να μα πείτε τι, προ, τι και αποτροπή έχει προβλέψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να μην υπάρξουν περαιτέρω χειραγωγήσει από την πλευρά των ε, αυτοκινητοπαραγωγών. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριο Ζωρίνιου. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Δεν θα είχε χρειαστεί να ζήσουμε τόσα σκάνδαλα αν υπήρχαν οι ανάλογες πρακτικές και δοκιμές για τον ελέγχο των εκπομπών. Καλώ λοιπόν έγινε προτεραιότητα να έχουμε καθαρά οχήματα τώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για του πολίτε, για την υγεία του και για να επιτύχουμε του στόχου μα για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Σημαντικό είναι να έχουμε φιλόδοξου στόχου, αλλά ακόμη πιο σημαντικό είναι στην πραγματικότητα να επιτευχθούν και στην πράξη. Διότι εγώ προτιμάω να μην μιλάω για φιλοδοξία στόχων, αλλά για φιλοδοξία στην υλοποίηση. Και για να υπάρξει αυτή η υλοποίηση είναι σημαντικό, για παράδειγμα, να υπάρξει συσχετισμό όλη αυτή τη διαδικασία και ενό νέου πλαισίου έρευνα για το νέο ε, κύκλο δοκιμών. Εδώ θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα υπάρχει η κατάλληλη κινητοποίηση στην έρευνα και την καινοτομία, στην έρευνα και την ε, ασφάλεια. Επίτροπε, νομίζω λοιπόν ότι θα χρειαστεί ένα νέο πλαίσιο ε, στην ε, ανάπτυξη των δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις. Και Καλό θα ήταν να παραμείνει αμετάβλητη αυτή η φιλοδοξία για να είμαστε πρωταγωνιστές στη μετάβαση σε καθερότερα οχήματα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία Λουκατσεύσκα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πιστεύω ότι η επιτυχία δεν είναι κάτι που θα εξαρτηθεί μόνο από τους πολύ φιλόδοξους στόχους. Κυρίως το θέμα είναι αν αυτοί οι στόχοι θα επιτεθούν. Μιλάμε για καθαρά οχήματα, μιλάμε για ηλεκτροκίνητα οχήματα. Έχουμε πολλά προβλήματα όμως ακόμα μπροστά μας, διότι το πρόβλημα θα είναι και η τιμή, το κόστος. Το θέμα είναι αν οι καταναλωτές θα αγοράζουν αυτά τα οχήματα, αν ε, έχουν μια προσιτή τιμή, ε, αν θα μπορούν να, τα, να επιτρέψουν στον εαυτό τους να τα αγοράσουν, αν θα μπορούν να τα φορτίσουν, αν θα υπάρξουν υποδομές επαναφόρτησης, ε, αν θα ταξιδεύουν μόνο με 100 χιλιόμετρα αυτονομίας ή αν θα υπάρξει μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας. Εδώ λοιπόν ένα πρόβλημα που έχει τεθεί εδώ και στην Επιτροπή Μεταφορών. Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα έχουν ανάγκη από λίθιο και κοβάλτιο στην παραγωγή του. Τα σπάνια αυτά μέταλλα εξορίσσονται στη Ζάμπια, στο Κονγκό, στη Χιλή, στη Λατινική Αμερική γενικότερα. Ήθελα να μου πείτε αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει κάποια μελέτη ή ανάλυση για τα αποθέματα αυτών των σπάνιων μετάλλων, για τη δυνατότητα διαρκούς ανεφοθιασμού σε πρώτε ύλε όπω αυτέ. Διότι τα μετάλλα αυτά εξορίσσονται σε χώρε που πολιτικά είναι σταθεί. Αυτό δεν θα θέσει να αμφιβόλο την όλη μας, το όλο μα εγχείρημα για τα ρητοκίνητα οχήματα. Ευχαριστούμε και η κυρία Γιάλα Σέντερ τώρα. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ να ευχηθώ καλή ανάρρωση στον Επίτροπο για το χέρι του. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με αυτά που σχόλησαν και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, αν δηλαδή θα είναι δυνατόν το συντομότερο δυνατό να έχουμε μια ανάλυση όσο το πιο λεπτομερή για τον κύκλο ζωής όλων των συστημάτων δηλαδή βενζίνη, υδρογόνο, ντίζελ, ρεύμα κτλ για να κάνουμε μια σύγκριση για την παραβολή του κύκλου ζωής. Γιατί μας έρχονται διαφορετικές και ε, αμφι... μεταξύ τους πληροφορίες. Το δεύτερο από τις προτάσεις σας, βλέπω ότι το ΣΕΦ, το Connecting Europe Facility, είναι ουσιαστικά για πολλά μέτρα το, ε, ο κορβανάς από τον οποίο παίρνετε τα χρήματα. Εγώ πιστεύω ότι ακριβώς θα πρέπει εδώ να κάνουμε τη διαφορά. Έχουμε αυτό το μέτρο, ε, το CEF, για να έχουμε ένα μετασχηματισμό του συστήματος ε, τα τελευταία ε, επόμενα χρόνια, τα επτά επόμενα χρόνια για την κινητικότητα. Στις συστάσεις του εξαμήνου θα μπορούσατε με αντικυκλικά μέτρα ίσως γιατί αυτό φαίνεται να λέει η πιθανή συμφωνία στη Γερμανία. Ο Επίτροπο Έτιγκερ αυτό φαίνεται να θέλει να προτείνει. Αν υπάρχει λοιπόν αυτή η δυνατή, δυνατότητα να δώσουμε αυτά τα κίνητρα. Επίσης 12 εκατομμύρια θέσεις εργασίας λέτε 4 για τις μπαταρίες. Έχετε ένα χρονοδιάγραμμα. Στα κράτη-μέλη προετοιμάζονται. Πώς θα εκπαιδευτεί αυτός ο κόσμος. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, αυτές ήταν οι ερωτήσεις. Έχετε τώρα το λόγο να απαντήσετε. Ας προσπαθήσουμε να δώσουμε λίγο προοπτική σε ορισμένε από τις ερωτήσεις, να εξήγησουμε κάποια πράγματα. Κυρίως διότι κάποιοι από εσάς μιλήσατε όχι μόνο για το στόχο του 40% που συζητήσαμε προηγουμένως, αλλά προσθέσετε και άλλο ένα στοιχείο στους στόχους του 2040 και στην ενεργειακή κατάσταση εκείνη την περίοδο. Τι ήθελα να πω τώρα. Το πλαίσιο που έχουμε στο χρονοδιάγραμμα έχει οριζόντα το 2030. Αυτό αφορά όλες τις προτάσεις μας, το σύστημα εμπορίας εκπομπών, τον επιμερισμό των προσπαθειών, το LULUCF, τους στόχους ε, διοξιδίου του άνθρακα, για τα οχήματα και για τα ελαφρά φορτηγά στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχουμε βάσει τη Συμφωνία του Παρισιού. Τουλάχιστον 40% περικοπή των εκπομπών μέχρι το 2030 και όλη μας η νομοθεσία είναι εστιασμένη σε αυτό το στόχο, σε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Τοπικά τώρα είναι βέβαιο ότι θα πρέπει να εξετάσουμε όλους τους ε, τομείς για να δούμε τι θα γίνει με την στρατηγική ε, απαλλαγή από τις 400 εκπομπές, ε, στο θέμα, να δούμε το θέμα διακυβέρνησης και τα ενεργειακά σχέδια και τα σχέδια δράση για το κλίμα και οι μακροχρόνιες στρατηγικές των κρατών μελών πρέπει να περιλαμβάνουν όλα αυτά τα στοιχεία. Αυτό ήθελα να ξεκαθαρίσω. Το δεύτερο είναι ότι αυτή η πρόταση έχει περιορισμένο εύρο όσον αφορά το διοξίδιο του άνθρακα. Δεν μιλάμε για τα οξίδια του αζότου ή τα μικροσωματίδια. Εγώ υποστηρίζω τις πολιτικές του Επιτροπού Βέλα και της Επιτροπού Μπιενκόφσκα στου τομείς αυτού. Τέθηκε το ερώτημα του κατά πόσο ε, ποιος ακριβώς ευθύνεται, όποτε έχουμε μεγάλη υπηρεκτικότητα σωματιδίων, πρέπει να δράσουμε σε όλα τα κράτη-μέλη. Στα κράτη-μέλη διαφέρουν οι ευθύνες. Αλλού είναι η κυβέρνηση, αλλού είναι άλλες αρχές της μεγάλες πόλεις, ε, οι Δήμοι των Πόλεων έχουν την ευθύνη να λάβουν οποιαδήποτε μέτρα είναι δυνατόν για να διασφαλίσουν την ποιότητα του αέρα για τους πολίτες και να διασφαλίσουν την υγεία των πολιτών. Τώρα εδώ αυτό που έχουμε το ο φάκελος αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα αλλά δεν αφορά μόνο το διοξιδίο του άνθρακα όπως ξεκίνησε περιλαμβάνει και μια συνιστόσα ηλεκτροκίνησης για τα ε, οχήματα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών. Αυτό προστίθεται στο πακέτο αυτό και εδώ έχουμε μια ανοιχτή συζήτηση και θα δούμε ποιο είναι το επίπεδο φιλοδοξίας. Έχω συνηθίσει το Κοινοβούλιο να κάνει ε, ε, φιλόδοξες προτάσεις. Αλλά με την ηλεκτροκίνηση αυτό που με ανησυχεί κυρίως είναι η έλλειψη υποδομών και πολιτικής βούλησης για φιλοδοξίες προτάσεις. Εγώ μάχομαι εντός της Κομισιόν και στους τριμερείς διαλόγους και παντού για αυτό στους σκοπούς. Και τώρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και άλλα στοιχεία. Τα αναλλακτικά καύσιμα, την οδηγία για τα αναλλακτικά καύσιμα. Πρέπει να προσπαθήσουμε να λειτουργήσουμε με τα ταμεία που έχουμε, με τις πολιτικές που έχουμε, να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε ε, μέσο έχουμε για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα υποδομής. Θα κάνει η Κομισιόν ό,τι μπορεί για το εγχείρημα αυτό. Τώρα το τελικό προϊόν, ξέρετε, δεν μας είναι άγνωστο. Κάποιοι είχαν πει, ε, κάποιος είπε εδώ να καλέσουμε κόσμο εδώ και κάποια μεγάλα ονόματα. Να ξέρετε ότι όταν εκπονήσαμε την πρόταση, συμβουλευτήκαμε τους πάντες. Και σίγουρα όλα τα λόμπι με απόλυτη διαφάνεια. Συμβουλευτήκαμε όλα τα λόμπι, όλο τον κόσμο, τους πάντες, τα συνδικάτα. Πρέπει να ακούσουμε, να εισακουστούν και αυτά. Τι θα γίνει με την ε, αλλαγή των δεξιοτήτων που χρειαζόμαστε για να τροποποιήσουμε τον τομέα, διότι θα φύγουμε από την καύση, από τις τεχνολογίες καύσης. αλλά δεν έχουμε γνώσεις για μπαταρίες και ηλεκτροκίνηση. Έχουμε μηχανικούς, έχουμε τις δυνατότητες, αλλά πρέπει να επανεκπαιδεύσουμε ολόκληρο το εργατικό δυναμικό μας. Και αυτή τη διαδικασία πρέπει να τη διαχειριστούμε έξυπνα, διότι οι τομείς αυτοί εξακολουθούν να είναι σημαντικοί προς όφελος των καταναλωτών, αλλά και προς όφελος των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών. Κύριε Τούρμες, λοιπόν, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αυτό είναι βέβαιο, να είστε βέβαιο. Αλλά ξέρετε, και εγώ το σκέφτηκα πολλές φορές, έχω περάσει από όλα τα έγγραφα διαβούλευση που μπορείτε να φανταστείτε. Έχω διαβάσει τα πάντα, έχω διαβάσει για όλες τις τεχνολογίες και για μένα η πρόταση αυτή είναι αρκετά ισορροπημένη. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, αλλά η αρχιτεκτονική, ξέρετε, έτσι είναι οι ισορροπημένε ε, προτάσεις τελικά. Πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλες τις συνέπειε ε, για όλα τα κράτη-μέλη, για όλους του ενδιαφερομένους, πώς επηρεάζουν τα πάντα, τις διάφορες επικράτειες. Σίγουρα η πρόταση αυτή αφορά μέχρι το 2030 και θα έρθει πολύ γρήγορα το 2030. Τα πράγματα αλλάζουν ταχύτατα. Είδαμε τι γίνεται με τα ηλεκτρικά ποδήλατα, με τα ηλεκτρικά οχήματα, βλέπουμε τις εξελίξεις της πόλης μας. Και μετά τίθεται και το θέμα των μπαταριών. Αυτό είναι Βέβαια Συζητάμε, λέμε τι θα γίνει με τι μπαταρίε. Ε, ε, κοβάλτιο, λίθιο, τι θα γίνει με το Κονγκό. Μιλάμε για μπαταρίε πρώτη γενιά. Τι θα γίνει μετά με το γραφένιο, με το υγρό γραφένιο στο μέλλον. για τις νέες μπαταρίες για το μέλλον. Εκεί θα μπορούσε να ηγηθεί η Ευρώπη των τεχνολογιών. Και τι θα γίνει τώρα με, την, με τις ε, παραγωγές μεγάλης κλίμακας στην Κίνα. Χρειαζόμαστε τεχνολογία για να μεταφέρουμε την παραγωγή εδώ. Και το ίδιο ισχύει και για τα ηλεκτρικά οχήματα. Το πρόβλημα που είχα είναι ότι δεν υπάρχουν υποδομές αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν εργαλεία. θα έχουμε ε, το σύστημα εξυπηρέτησης κατά προτεραιότητα και θα χρησιμοποιήσουμε και τα διαρθρωτικά ταμεία. Κυρία Γιώσο. γιατί τη μάζα που αναφέρατε έχουν, ε, υπάρχουν διάφορες επιλογές ε, έχουμε τις παραμέτρους μάζας ε, της ωφέλειας όλα αυτά έχουν συμπεριληφθεί στους ίδιους στόχους για όλους τους κατασκευαστές η προσέγγιση μάζας είναι η απλούστερη που θα καθορίσει τις μελλοντικές προσπάθειες των αυτοκινητοβιομηχανιών. Αν αλλάξουμε ε, προσέγγιση ε, τα πράγματα είναι απρόβλεπτα. Η πρόταση προβλέπει προσαρμογή της μάζας αναφοράς που αναφέρεται στη μάζα του στόλου αυτοκινήτων ως κίνητρο ε, ώστε να υπάρχει κίνητρο να αποφύγουμε την αύξηση της μάζας. Το μερίδιο των ηλεκτρικών οχημάτων που θα κυκλοφορούν θα καταστήσουν λιγότερο σημαντική την παράμετρο της ωφέλειας. Αυτά όσον αφορά τις εκπομπές. Επειδή ζητήσατε να μιλάμε για διαφάνεια, ε, η απόφαση παρακολουθήσης ενημερώνει για τις αποφάσεις ε, περί διοξιδίου του άνθρακα των κατασκευαστών και για τα πρόστιμα. Ακούσαμε μια ερώτηση γιατί δεν λαμβάνουμε υπόψη κατά πολέμηση των ε, εκπομπών την προσέγγιση κύκλου ζωής και το είπαν και άλλοι νομίζω αυτό. Η εκτίμηση αντικτύπου υπογραμμίζει την πρόταση επιλογής ε, ε, για να λαμβάνονται υπόψη οι νέοι στόχοι του άνθρακα. Βάσει τη αξιολόγηση κύκλου ζωή θα είχαμε διπλού κανονισμού και θα δημιουργείται σύγχυση όσον αφορά τι ευθύνε ε, και τη λογοδοσία. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες ε, θα αποκτούσαν ευθύνε για εκπομπέ που λαμβάνουν χώρα εκτός του τομέα. Μια τέτοια διαδικασία υπάρχει κίνδυνο επίση να δημιουργήσει επιπλέον φόρτο, ειδικότερα ε, σε θέματα παρακολούθησης και υποχρεώσεων. η εστίαση στι εκπομπέ ε, διοξιδίου του άνθρακα στι αυτοκινητοβιομηχανίε συνάδει με άλλε πολιτικέ ε, που σχετίζονται με την κλιματική πολιτική τη Ένωση και για το σύστημα εμπορία εκπομπών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τις διάφορες πρωτοβουλίες. Ε, τώρα όσον αφορά τα βιοκαύσιμα έχουμε βασίσει την προσέγγιση μας στην σαφή ευθύνη για σαφείς ε, φορείς ε, η νομοθεσία αυτή εφαρμόζεται απευθείας στους κατασκευαστές αυτοκινήτων που δεν μπορούν να ελέγξουν πώς θα χρησιμοποιηθούν τα αυτοκίνητά τους. Τα ίδια αυτοκίνητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με κανονικά καύσιμα ή με βιοκαύσιμα εμείς έχουμε αποφασίσει ε, να ακολουθήσουμε την προσέγγιση ε, tailpipe, ε, την προσέγγιση των εκπομπών, το οποίο λαμβάνεται υπόψη και σε άλλα νομοθετήματα. Τα βιοκαύσιμα υπάρχουν στη νέα οδηγία όπου έχουμε συμπεριλάβει μια εντολή για τους προμηθευτές καυσίμων μέχρι το 2030 να περιλαμβάνουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό βιοκαυσίμων στην αγορά. Διάφορα νομοθετήματα δηλαδή ε, συμβάλλουν στην όλη κατάσταση ε, αποφεύγοντας τη διπλή νομοθεσία και κατανέμοντας ε, ευθύνες. Υπήρξε και μια ερώτηση από την κυρία Μάισνερ που μας λέει γιατί να αναπτύξουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα όλο το ηλεκτρικό ρεύμα δεν παράγεται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και το ερώτημα που τίθεται είναι Συμβάλλουν πραγματικά τα ηλεκτρικά οχήματα στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα στον κύκλο οδήγηση, στον κύκλο ζωή του. Το πρώτο πρέπει να πούμε ότι οι εκπομπέ αερίων θερμοκηπίου από αυτό το τομέα μειώνονται ταχύτερα από ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο τομέα. Στον τομέα αυτό του παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματο μειώνονται. Και με τι προτινόμενε πολιτικέ, ε, το αναθεωρημένο ETS και η αναθεωρημένη οδηγία για την ενέργεια ε, καθιστά δυνατή την απαλλαγή από ανθρακούς εκπομπές μέχρι το 2030 της ηλεκτροπαραγωγής. Μέχρι τότε ε, ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής θα έχει μειώσει την παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου. Έχει μειωθεί λοιπόν, θα μειωθεί. Με τη νέα λοιπόν πρόταση υπάρχει και ένα στοιχείο που βασίστηκε στο ε, κοινό κέντρο έρευνα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δείχνει ότι τα αυτοκίνητα που κινούνται με μπαταρίε και σχετικέ λεπτέ πλάκε θα έχουν χαμηλότερε εκπομπέ και από και όταν συγκρίνουμε το τι παράγεται με, την, ε, με τα καύσιμα από την ηλεκτροκίνηση. Το 2030 ο μισός όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τις μπαταρίες ηλεκτροκινήτων και ο μέσο όρο εκπομπών μάλλον θα είναι 70-75% χαμηλότερος από τη, σε σχέση με τον diesel και τα πετρελαιοκίνητα. Ε, τα, οι μπαταρίε και οι λεπτέ πλάκε θα έχουν τουλάχιστον 55% διαφορά σε σχέση με τα πετρελαιοκίνητα. Ε, σε επίπεδο, τα βενζινοκίνητα μάλλον, σε σχέση με το τι συμβαίνει στα κράτη-μέλη μέχρι το 2030, για τις μπαταρίες και μόνο οι εκπομπές θα έχουν μειωθεί δραστικά σε 22 28 χώρες. Τώρα αυτό συμβαίνει μόνο σε έξι κράτη-μέλη. Επιπλέον, η ανάλυση της μελέτη αντικτύπου δίνει, δείχνει ότι η δίσδυση των ε, αυτοκινήτων ε, με μπαταρίες και τι μπαταρίες θα είναι χαμηλότερη σε κράτη-μέλη που το μείγμα των ε, χαμηλού άνθρακα και ηλεκτροκινήτων είναι μεγάλο. Αυτά, κυρία Πρόεδρε, για τις απαντήσεις στις ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής ΕΝΒΗ. να πω και στη συνεργασία των ε, μελών σας για να βελτιώσουμε αυτή την πρόταση νομοθεσίας και ελπίζω ότι θα προκύψει ισχυρή από το Κοινοβούλιο για να περάσουμε στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο που θα είναι καθοριστικής σημασίας. Αυτά τα τόσο σημαντικά ε, θέματα και κανόνες που θα μας επιτρέψουν να περιορίσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και να βελτιώσουμε την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα για τους πολίτες μας. Ευχαριστούμε, Επίτροπε. Υπάρχει, είδατε, μεγάλο ενδιαφέρον για αυτή την νομοθετική πρόταση. Περιμένουμε και η κυρία Ντάλι να ξεκινήσει. Ε, ευχαριστούμε πολύ. Συνάδελφοι, σα ευχαριστώ πολύ όλου για τη συζήτηση. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε για να συνεχίσουμε παρακαλώ. Σήκωση, 21 γλώσσες διερμηνία και έχετε ηλεκτρονικά το φάκελο μέσω του e-meeting. Επίσης, για τα διοργανικά θέματα, διοργανικές διαπραγματεύσει. Δεν ξέρω καν χρειάζεται να σας την συστήσω. Σας καλέσαμε εδώ να μας κάνετε μια παρουσίαση. Πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. σας ευχαριστώ που με καλέσετε σήμερα στην ετησιακή ανταλλαγή απόψεων. Είναι η πρώτη ετήσια κράση ως διευθύντριας ε, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Έλεγχου Νόσων, η CDC. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνεχή δέσμευσή σας. Θέσατε πρόταση ψηφίσματος για να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τους εμβολιασμού. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Καταρίνα Κονέτσινα που είναι ο σύνδεσμος και πάντοτε υποστηρίζει την την υπηρεσία μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους σε τι κάναμε το 2017 και τι σκοπεύουμε να κάνουμε το 2018 ως προτεραιότητα. Η αντίσταση στα αντιμικροβιακά φάρμακα. Αυτό είναι εστίασή μας και αυτό είναι επίκεντρο για τις δράσεις μας και στο μέλλον. Θέλουμε να μειώσουμε και την μικροβίων όπως το πένεμα, εντερομπακτεριακέ. Για τα εντεροβακτηρίδια θα απαιτηθούν περισσότερα ε, δημοσιοποιήσει δύο έγγραφα. Πρώτον, την έκθεση ε, την τζαϊάκρα όπως λέγεται για την αντιμικροβιακή κατανάλωση και αντοχή και επίσης την Κοινή Επιστημονική Επιτροπή για κάποιους δείκτες φαρμάκων στον άνθρωπο αλλά και στα ζώα που παράγουν ε, τρόφιμα. Πάντα σε συνδυασμό με την ΕΦΣΑ και τον EMA. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το 2018 την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την ε, εφαρμογή του άρθρου ε, One Health Action λα. Στα κράτη-μέλη, ξεκινήσαμε ήδη από την προηγούμενη χρονιά. Επίσης, ε, θα κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις ότι αφορά το φόρτο, το βάρος ε, της ε, μικροδιακής αντοχής και θα μιλήσουμε και για κάποιες μελέτες εντατικής φροντίδας και σε άλλες εγκαταστάσεις. στη διάρκεια του έτους. Το ίδιο θα κάνουμε και το 2018. Να τονίσω κάποιες από τις δραστηριότητες για τη βελτίωση της κάλυψης και την αντιμετώπιση αυτού του δισταγμού για τον εμβολιασμό. Ένα παράδειγμα είναι ότι έχω σε ό,τι αφορά την πληροφόρηση που δίνουμε για τα εμβόλια. Πέρυσι είχαμε και ένα ευρωπαϊκό φόρουμ υγείας. Εκεί οργανώσαμε ένα workshop για να αντιμετωπίσουμε το δισταγμό των ανθρώπων να εμβολιαστούν. Τονίσαμε πόσο πολύπλοκο είναι αυτό το φαινόμενο και είπαμε ότι πρέπει να περάσουμε από την τώρα έχουμε την εβδομάδα ανοσοποίησης τον Απρίλιο. Θα έχουμε λοιπόν μία ανακοίνωση και μία εργαλειοθήκη για τα κοινωνικά μέσα δικτύωση, για να καταπολεμηθεί ακριβώς ο δισταγμός, να βοηθήσουμε τα κρατη και επίσης ε, σε ό,τι αφορά τις ε, διάφορες νόσους, ε, στοιχεία για για το φόρτο, για το βάρος ορισμένων νόσων και ιδίως για την ερυθρά. Έχουμε επίσης έγγραφα ε, που θα δημοσιοποιήσουμε για τον ε, ε, ιό HPV, το ανθρωπίνο θυλώματος και για τα αγόρια αυτού του ιού. Επίσης υπάρχουν και άλλες νόσοι που θα παραμείνουν ψηλά στη διάταξη όπως είναι η φυματίωση. Θέλουμε να τηρήσουμε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Θα πρέπει λοιπόν για της, ε, για την φυματίωση ε, την νόσο αυτή, θα έχουμε δε και την πρώτη ψηλού επίπεδου συνάντηση στο πλαίσιο του ΟΗΕ για την ε, φυματίωση την νόσος, υπατήτηδα. Θέλουμε ε, να έχουμε ένα πρόγραμμα παρακολούθησης της νόσου μαζί με το αρμόδιο οργανισμό και σημάτων. Εμείς παρακολουθούμε επικαθημερινής βάσεως τις νέες απειλές για την υγεία που θα μπορούσαν να προκύψουν. Είχαμε δύο αξιολογήσεις ε, φέτος για τη Σαλμονέλα Αγκώνα και για τον κίτρινο πυρτό στην ε, Βραζιλία. Και βλέπετε εδώ τις μελλοντικές τεχνολογίες για το έργο μου. Έχουμε την αλληλεγγύα του γονιδιώματος, αλληλεγγύη του γονιδιώματος. Ε, που μας βοηθάει στις προειδοποίησεις και θα στηρίξουμε και την τεχνολογία της e-health, της ηλεκτρονικής υγείας για την επιτήρηση νόσων και την αξιολόγηση κινδύνων. Το 2000-2017 ε, συνεχίσαμε να ενισχύουμε την τεχνική μας συνεργασία με πρωτοβουλίες επίσης δημιουργίας δυνατοτήτων το μέλλον τώρα. Θέλουμε να δούμε τι θα κάνουμε τον προπολογισμό μας. Είχαμε πέρυσι 58 εκατομμύρια και όπως βλέπετε 99,8% τα έχουμε ε, δεσμεύσει και ήδη το 81% το έχουμε εκταμιεύσει. Αυτό και αυτή η ορεινή περιοχή ε, σημαίνει ότι ποια είναι αυτά τα ποσά που γύρισαν πίσω φέτος ε, είναι πάρα πολύ λίγα τα... αυτό το βουνό όπως φαίνεται. Τέλος πάντων αυτό το διάγραμμα δείχνει πόσο είμαστε στην κάτω. λίγο θα εγκαινιαστεί η νέα αυτή ε, εγκατάσταση. Ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεστε εδώ, που βρεθήκατε εδώ. Έχουμε πολλούς συναδέλφους που θέλουν να πάρουν το λόγο. θα δώσω το λόγο στην κυρία Κονέτσνα για την η επαφή μας με την ECDC. Την e Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιό την κυρία Διευθύντρια, σας καλωσορίζω. Είναι εδώ και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από πλευράς Κοινοβουλίου. μας δώσετε εσείς, γιατί είστε παρούσα σε όλες τις συζητήσεις, σε μια νέα ματιά. Φέτος, είτε σπον τον ελπίζω, επίσης ε, να μετακομίσετε ομαλά, είναι σχεδόν καινούργιο αυτό το κτίριο και εκεί που θα πάτε λοιπόν ελπίζω να μπορέσετε να κάνετε και καλύτερα τη δουλειά σας, να υπάρχει καλύτερα συντόνιση έργο σας πολύ καλύτερα. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήρε αυτή την απόφαση για τη μετακόμιση αυτή. Δεν ήταν δυνατόν ε, να ε, συνεχίσετε να δουλεύετε σε ένα τέτοιο περιβάλλον όπως μέχρι πριν τις ε, άλλες δύο που αναφέρατε. Ουσιαστικά η Κομισιόν διστάζει να πάρει πρωτοβουλίες. Και ουσιαστικά από εσά μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες για αυτές τις ε, τρει νόσους, AIDS ε, και φυματίωση. Είναι όμως πάρα πολύ ε, σημαντικά αυτά τα θέματα. Πολέμηση αυτών των τριών νόσων. Σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό έχω μια ερώτηση. Σας ευχαριστώ που αναφέρατε το θέμα αυτό και σας ευχαριστώ που ασχολείστε με το θέμα αυτό. Οι δικοί σας κάθε μέρα έχουν αντιμετωπίσουν κάποιους μύθους που μου μιλήσατε για κάποια project στην Αυστρία και στην Ιταλία το 2017. Πότε, μάλλον ήταν καλά αυτά τα ε, σχέδια, θα ήθελα να μου πείτε, είχαν ε, καλά αποτελέσματα. Θα μπορούσαν να υιοθετηθούν αντίστοιχα και σε άλλες χώρες. Η Ιταλία έχει μεγάλο πρόβλημα με την Ιθρά, αλλά όχι μόνο, υπάρχουν και σε άλλες χώρες όπως η Γερμανία αντίστοιχα προβλήματα. Θα ήθελα να μειώνονται τα ποσοστά των μεταδοτικών αυτών ασθενειών στην Ευρώπη. Αυτό εύχομαι. Και σίγουρα πρέπει να σας αποσχολήσει το θέμα και στο μέλλον με την ίδια προσοχή. Σας ευχαριστώ επίσης για όσα κάνετε και για την ε, μικροβιακή αντοχή. Κρίμα που δεν καταφέραμε να πιέσουμε την ε, βιομηχανία να ασχοληθεί με το θέμα αυτό που η φαρμακοβιομηχανία δεν φαίνεται αντιλαμβάνεται το πρόβλημα. Υπάρχει κίνδυνος όμως. Δηλαδή υπάρχει κίνδυνος να χάσουν τη ζωή τους ασθενείς από συνηθισμένες αρρώστιες λόγω της αντοχής που είναι και τόσο ευρέως διαδεδομένη ώστε τα κανονικά φάρμακα τελικά να μην έχουν ε, δράση σε κανέναν. Ξέρω ότι η δική σας βασική ε, δραστηριότητα, το βασικό σας καθήκον να μας ενημερώνετε βέβαια εδώ, αλλά νομίζω ότι και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να σας απασχολήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κονέτσνα. Δίνω το λόγο τώρα στα μέλη που είπαν ότι θέλουν να μιλήσουν. Κυρία Ριβάζη, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλωσορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γνώριζα την προκατοχό σας. Ε, διότι είστε αρμόδια για τις μολυσματικές ασθένειες. Πώς να μπορεί να προβλέψει κανείς τέτοιου είδους ασθένειες, αυτό είναι το ερώτημα. Μιλήσατε πολύ για τον εμβολιασμό. Πώς να μπορεί να προβλέψει κανείς τέτοιου είδους ασθένειες, αυτό είναι το ερώτημα. Μιλήσατε πολύ για τον εμβολιασμό, 42% ανθρώπων οι οποίοι διστάζουν να εμβολιαστούν. Και πρέπει να ρωτηθούμε γιατί. Γιατί τέτοια αντίσταση. Λέει ότι πρέπει να εμβολιαστούν. Γιατί, διότι υπήρξαν πολλές συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των εμπειρογνωμόνων που ήταν αρμόδιοι στο τεχνικό κέντρο και με, την, ε, με το εμβόλιο κατά της... Ε, και με τη γρήπη HN1 είχαν υπάρξει αυτά τα θέματα που έκαναν τους ανθρώπους καχύποπτους. Στην Γαλλία τώρα λοιπόν λέμε ότι υπάρχει υποχρέωση εμβολιασμού και και υπάρχει εξαιρετική κάλυψη διότι ο κόσμος ε, έχει εμπιστοσύνη στις αρχές. Για μένα λοιπόν δεν είναι υποχρέωση που θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, υπάρχουν πολλά αιτήματα όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός ε, Υγείας λέει ότι πρέπει να Παλιότερα ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας έρεγε 70% και μετά πήγαν στο 80% και τώρα είναι 95%. Ποια επιστημονική μελέτη το αποδεικνύει αυτό. Δεύτερον, σε επίπεδο εμβολιασμού για πολύ καιρό στη Γαλλία κάναμε διάφορα εμβόλια για διάφορες ε, ασθένειες. Μπορείτε να κάνετε λοιπόν μελέτες κόστους οφέλους για κάθε εμβόλιο για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη. Πολλέ αμφιβολίε υπάρχουν για τις πρόσθετες ουσίες, συστατικές ε, ουσίε που υπάρχουν μέσα. Ε, τον προκατοχό σα για την αρκοληψία. Ξέρετε, είχαμε ένα εμβόλιο που είχε δημιουργήσει κάποια προβλήματα στη Σουηδία και στη Φιλανδία. Και τελευταίο σκάνδαλο και θέλω να μου πείτε τι γίνεται με αυτό για τον δάγκιο πυρετό. Ξέρετε, είχαν εμβολιαστεί 700.000 παιδιά. Όλα αυτά τα σκάνδαλα ο κόσμος είναι καχύποπτος όσον αφορά τον εμβολιασμό. Τι μπορείτε λοιπόν να μας πείτε ε, για αυτό το εμβόλιο κατά του δάγκιου πυρετού. Εγώ ζήτησα τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, δεν έχει ακόμα δώσει την άδεια, αλλά όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά δημιουργούν αυτή την αντίσταση. Ευχαριστώ. Κέντρο ε, για την παρουσίαση αλλά και για την καλή συνεργασία για τα πιο διαφορετικά μεταξύ τους ζητήματα. Υπάρχει και έκθεση ε, πρωτοβουλίας από το Κοινοβούλιο για την Κροβική Αντοχή. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την καλή αυτή δουλειά, κυρίως γιατί είμαι αρμόδια στην Επιτροπή έμφυς προηγούμενες χρονιές, ότι έχετε λάβει υπόψη σα ε, τι προτρύνσεις της ε, επιτροπή μας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν ε, ανάγκες ε, βελτίωσης και προσαρμογή Σε αισθητική σας περίπτωση σε εξέλιξη είναι στο pipeline. Τώρα σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό. Είπατε ότι υπάρχει αυτή η καμπύλη προς τα κάτω. Θεωρείτε ότι έχετε επαρκή ε, προϋπολογισμό τα επόμενα χρόνια για να αντιμετωπίσετε τα αυξανόμενα καθήκοντά σας ή σε ό,τι αφορά το workload, το, βάρτο, το φόρτο εργασίας, θεωρείτε ότι έχετε επαρκή στελέχωση και έχετε και επαρκή προπολογισμό, επαναλαμβάνω, φέρετε πέρα και ένα άλλο ε, ένα κοπλιμέντο, αν θέλετε, για την πληροφόρηση, τη διαφάνεια. Πάρα πολύ θετικό. Και δεν είναι απευθύνεται μόνο σε εμπειρογνώμονες, αλλά και στον μέσο καταναλωτή, αν μπορώ να το πω έτσι που βλέπει αυτά τα πάρα πολύ ευανάγνωστα και εύκολα κατανοητά διαγράμματα και άλλα σχήματα, ώστε να... Να ε, τα ευχαριστώ. Κύριε Μάισνερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και Κύψουν. Εγώ νομίζω ότι είναι κάτι ε, σημαντικό. Πρέπει πάντοτε να το έχουμε υπόψη. Το Νοέμβριο μιλήσετε για μια δημοσίευση και επί Ολλανδικής Προεδρίας το θέμα ήταν προτεραιότητα αυτό το θέμα. Όχι και τόσο πια για τις επόμενες παιδίες, αλλά η ερώτηση μου είναι η εξής, ε, η ολχής. Ε, πώς αντιδρούν ε, οι κλινικές, υπάρχει ανταλλαγή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι εθνική πολιτική υγείας, αλλά δεν υπάρχει ανταλλαγή βελτιστών πρακτικών σε αυτή την περίπτωση. Τι εμπειρία έχετε εσείς δεν ξέρω αν το περιλαμβάνει αυτό και η έκθεσή σα, θα είδαμε Ευχαριστούμε. Ο κύριος Πότς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τη δουλειά σας. Απλώς θα ήθελα να... Η κυρία Μάζεκ Κουκόβιτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ζητήσω συγγνώμη για την καθυστερήσή μου, διότι είχε φοβερή καθυστερήση η πτήση από τη Σλοβενία σήμερα. Να πω κάτι που ήταν τελείως σαφές κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, διότι δεν άκουσα την παρουσίαση. Απλώς να πω ότι το να εργάζεται κανείς στο Διοικητικό Συμβούλιο του ECDC είναι δουλειά που διέπεται από απόλυτη διαφάνεια. Και γι' αυτό οφείλουμε ευχαριστήσεις όχι μόνο στους διευθυντές, αλλά σε όλη την ομάδα. Η... Το υλικό που προετοιμάζουν είναι εξαιρετικό και βάσει αυτού εργαζόμαστε. Ίσως να πρόσθετα μερικά πράγματα. Υπό το φως των μελλοντικών εκλογών το 2019, είμαι βεβαία ότι τα αποτελέσματα που θα φέρει το κέντρο είναι απαραίτητα για να πείσουμε τους πολίτες ότι η προστιθέμενη αξία που προσφέρεται είναι όντως προστιθέμενη αξία. Χρειαζόμαστε λοιπόν όλοι κάποιους δείκτες που να ε, είναι αρκετά πιστικοί, ε, μερικά παραδείγματα ας πούμε για το πώς ε, το κέντρο πρόληψης και ελέγχου των νόσων ασχολείται με τις ανισότητες ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς ή ποια ήταν αυτή η συνεισφορά του κέντρου που έκανε τη διαφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ποιο βαθμό το κέντρο αποφεύγει την επανάληψη των ίδιων προσπάθειών των κρατών μελών, των διαφόρων οργανισμών και του ίδιου του κέντρου. Επίσης, πώς οι επιστήμονες ενισχύουν την προστασία της υγείας των πολιτών της Ένωσης από ενδεχόμενες απειλές της δημόσιας υγείας. Είμαι πεπισμένη ότι θα υπάρξουν πολλές θετικές επιπτώσεις και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες και θα ήταν πολύ πιο θετική αν ήξεραν τα αποτελέσματα που επιτυγχάρει το κέντρο. Εάν υπήρχε κάποιος που μπορούσε από το Ευρωκοινοβούλιο ας πούμε να εξηγεί και να προβάλλει στα κράτη-μέλη τι κάνουμε διότι με το Brexit σήμερα και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι πιο σημαντικό να γνωρίζουμε πώς θα αποδείξουμε την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στους πολίτες. Ευχαριστήσω την Αντρέα Αμών για τις προσπάθειές της και να την συγχαρώ για όσα κάνει για το πνεύμα. Συμφωνώ απολύτως με την συνάδελφο. Έτσι δουλεύουμε στο διοικητικό. Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι πραγματικά νομίζω χρειαζόμαστε περισσότερη ε, διάδραση και επικοινωνία με το Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό είναι κάτι που χρειαζόμαστε διακαώς. Περισσότερο να ερχόμαστε μια στο τόσο για μια ακρόαση. Είμαστε ακόμη σε ένα σημείο όπου η αντίσταση στα αντιβιωτικά είναι μεγάλη απειλή για την Ευρώπη και παρά την πολύ σκληρή δουλειά του κέντρου δεν μπορούμε να λέμε ακόμα ότι έχουμε το να μην υπάρχει μια ε, εκστατεία ενημέρωση απευθεία από το κέντρο ελέγχου και πρόληψη των νόσων, αλλά να αφήνουμε του εθνικού φορεί να αναλαμβάνουν αυτή την ενημέρωση, δεν είναι τελικά τόσο παραγωγικό. Μια άμεση εκστατεία θα ήταν ίσω απονικών φορέων. Δεν έχει πάντα το ίδιο αποτέλεσμα στο κάθε ένα από τα κράτη-μέλη. Πιστεύω λοιπόν ότι μια άμεση εκστρατεία με τη βοήθεια του Ευρωκοινοβουλίου θα μπορούσε να μας βοηθήσει εξαιρετικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. η κυρία Μαγκίνες δεν με είχε ενημερώσει ε, για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 ή τέλος πάντων 27 συν Ηνωμένο Βασίλειο. Πώς θα επηρεαστείτε και τι μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε ως προς το σύστημα Αιγέρης Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Αμών. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για όλα τα συγχαρητήρια για τις φιλοφρονήσεις για τη δουλειά μας. Όπως υπόθηκε δεν είναι προσωπικά. Ε, μπορεί να απουσιάζουν και επίσης να μην έχουν και χρόνο να μας ακούσουν αυτή τη στιγμή, οπότε θα τα μεταβιβάσω. Ε, για τις ερωτήσεις σε σχέση με τα εμβόλια και την... Ε, ε επιφυλακτικότητα, τη τη προσέγγιση που υπάρχει σε σχέση με τα εμβόλια. Για την Αυστρία και την Ιταλία. Το θέμα είναι να βοηθήσουμε να προσαρμόσουν τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουμε σε ένα σύνολο μέτρων για να ενημερωθούν ε, οι επιφυλακτικές μερίδες του πληθυσμού, ιδίως οι στο εθνικό επίπεδο. Βρήκαμε ότι δεν υπάρχει καλή μετάφραση. Πρέπει να υπάρχει μετάφραση στο, στις εθνικές προϋποθέσεις, συνθήκες της κάθε χώρας. Τα πράγματα διαφέρουν μεταξύ των χωρών. Αυτό θα πρέπει να γίνει όχι μόνο για την Ιταλία και την Αυστρία όπως έγινε πέρσι. Ήδη έγινε γίνει ένα αριθμό χωρών και γίνεται κατόπιν δικού τους αιτήματο. Διότι μερικές χώρες ε, τα φροντίζουν μόνες τους φυσικά. Ε, αυτά για τα εμβόλια, για την κυρία Ριβαζή. Θέσατε πάρα πολλές ερωτήσεις για την επιφυλακτικότητα σε σχέση με τα εμβόλια. Το ζουμί στην όλη υπόθεση και απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις είναι η εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη ξανεμίστηκε. Η εμπιστοσύνη του κόσμου προς αυτούς που ε, ευαγγελίζονται τα εμβόλια ως λύση. Ε, και ακόμη και αυτούς που τα προωθούν, τους εργαζόμενους στον τομέα υγείας. Έχουμε Ακόμα και στον τομέα της πρόνοιας της ίδιας ε, μεγάλη επιφυλακτικότητα προς τα εμβόλια. Την καλλιεργούν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Βρήκαμε ότι η επιφυλακτικότητα προς τα εμβόλια δεν είναι κάτι που μπορούμε να επιλύσουμε με ένα ενιαίο μέτρο για όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει πραγματικά να μπούμε στις λεπτομέρειες της κάθε χώρας, να δούμε γιατί το κοινό διστάζει. Γιατί καμιά φορά είναι θέμα ε, βολής. Ε, Θεωρώ ότι είναι τόσο περιπλοκό να εμβολιαστούν που προτιμούν να μην το κάνουν. Ε, άλλοι έχουν ε, απορίες. Άλλοι δεν εμπιστεύονται τα εμβόλια. Είναι λοιπόν πραγματικά ε, διαφορετικές αποχρώσεις. Διαφορετική βαθμή επιφυλακτικότητας. Και βεβαίω μπορεί να εξαρτάται και από το τι είδου εμβόλια προσφέρονται. Δηλαδή, οι παράγοντες που καθορίζουν την επιφυλακτικότητα σε κάθε χώρα μπορεί να διαφέρουν τελείως για την Ερυθρά ακόμα και στην ίδια χώρα. Εδώ να τονίσω ότι πρόκειται για ένα θέμα εξαιρετικά περίπλοκο. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι με αυτά τα κουτιά εργαλείων όπως λέγονται, τα toolkit, να διευκολύνουμε τις χώρες να βελτιώσουν την πληροφόρηση του κοινού, ιδίως όσον είναι επιφυλακτική. Βεβαίως, μελετούμε τι προσεγγίσεις έχουν υιοθετηθεί σε χώρες όπως η Ιταλία και η Γαλλία, που επέβαλαν την υποχρεωτικότητα των εμβολίων, ενώ άλλε χώρε ακολουθούν διαφορετική προσέγγιση. Όπως για να είναι σημαντικό να πω ότι πάντοτε αναφέρεται ότι δεν λειτουργούν τον ίδιο τρόπο τα ίδια μέτρα στην κάθε χώρα. Όπω είπατε, οι οι εργαζόμενοι του τομέα υγεία μπορούν να επιλέξουν και να δουν τι μπορεί να είναι λύση για τη δική του την περίπτωση. Αυτό το έχουμε ήδη κάνει. Εγώ χάρη. Κανεί δεν σκεφτόταν ότι θα υπήρχε τέτοια αντίσταση στο ανάλογο εμβόλιο. Το κοιτάζουμε λοιπόν. έχουν διαφορετική συνάντηση ερυθρά. Είναι εξαιρετικά μεταδοτική. Γι' αυτό πρέπει να είναι οι παρενέργειες. Πρέπει να παρακολουθούμε τις παρενέργειες και να έχουμε μία ε, διαφοροποιημένη προσέγγιση. Η νομοθεσία επιτρέπει, ε, επιβάλλει στους παραγωγούς την υποχρέωση να παρακολουθήσουν το τι γίνεται και στην αγορά ε, μετά τον εμβολιασμό. Επίσης η κυρία Κοπά έθεσε ένα θέμα για την... Ε, πρέπει να προσαρμοστεί στην ε, εθνική κατάσταση, τις συνθήκες της κάθε χώρας. Δεν είμαι βεβαίω ότι θα είναι περιόν να το λάβει υπόψη. Βεβαίω η βιομηχανία είναι ε, σημαντικό εταίρο στην όλη διαδικασία, αλλά δεν είναι ο μόνο. Δεν μπορεί να το κάνουν μόνο τους οι εταιρείε αυτό. Όλοι πρέπει να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι και να δούμε τι θα κάνουμε για να ευαισθητοποιήσουμε για το θέμα. Είναι ένα τμήμα του στο τόπο μας αφιερωμένο τις συμβολές των 100 μελών. Εκεί μπορούν τα κάτι μέλη να βάλουν τις προσώπους των 100 μελών, όπου καλλιεργούμε αυτή την επικοινωνία. Επίσης, για τις τάσεις, για την, ε, για την ε, φαρμακευτική δράση ε, πρέπει να κρατήσει για πολύ καιρό η όλη προσπάθεια. Για την κλειψέλ, είναι η τελευταία γραμμή στο βακτήριο. Όταν υπάρχει αντίσταση σε αυτό, οι επιλογές είναι ελάχιστες. Το είδαμε, είναι η εξέλιξη στον προπολογισμό. Και αυτό είναι τι παραπάνω θα μπορούσαμε να κάναμε αν είχαμε παραπάνω πόρου. Τώρα, ε, στη συζήτηση για το μελλοντικό προπολογισμό, έχουμε αναφέρει σε ποιου τομεί θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα. Τα έχουμε πει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμω όλα θα εξαρτηθούν από το πώ θα πάνε οι συζητήσει. Οπότε, ό,τι μπορούμε, κάνουμε με αυτά που έχουμε. Αν είχαμε περισσότερα, θα κάναμε και περισσότερα, είναι σαφέ. Και το τελευταίο ήταν για το Brexit. Αυτό είναι κάτι το οποίο αρχίζει να είναι ως προοπτική στον οριζόντα για μας, βαρύνει, ρίχνει τη σκιά του πάνω στη δουλειά μας. Έχουμε πολλούς συνεργάτες από το Ηνωμένο Βασίλειο και ανησυχούν τι θα τους συμβεί. Παρακολουθούμε όλες τις διαπραγματεύσεις και είμαστε και σε επαφή με όλο το υπόλοιπο δίκτυο των οργανισμών, γιατί δεν θα επηρεαστεί μόνο το κέντρο μας. Αυτό που θα συμβεί, ε, η, η έκβαση των διαπραγματεύσεων, θα επηρεάσει συμβάσεις και συνεργασίες που έχουμε με το Ηνωμένο Βασίλειο, με δικούς τους φορείς, τι μπορούμε να κάνουμε μετά το Μάρτιο του 2019, αυτό θα επηρεαστεί επίσης, ε, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να το σεβαστούμε. Όποια λύση βρεθεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ισχύει και για μας. Ε, είναι σαφές ότι έχουμε συνεργασία και με χώρες εκτός Ένωσης για εντοπισμό κρουσμάτων, για έρευνα, για συνεργασία ερευνητική. Με τον ένα τον άλλο τρόπο θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να, κάνουμε το, να επιτρέψουμε τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου ανάλογα με το τι λύση θα έχει βρεθεί. Ελπίζω ότι απήντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Ναι, ναι, βεβαίως και απαντήσατε. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Μείνετε εδώ. briefly, uh, since I had to report back on you on uh, interinstitutional Έπρεπε να σας πω, γυρίζω στο προηγούμενο σημείο για τις οργανικές διαπραγματεύσεις πρόσφατα. Είχαμε δύο ζητήματα τα οποία μας απασχόλησαν. Το πρώτο ήταν για την ε, τροποποίηση του κανονισμού για την τριμερή διάλογο 21 Ιανουαρίου με τη Βουλγαρική Προεδρία. Καλύψαμε πτυχές ε, που αφορούσαν ε, τις θέσεις ε, Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για την πρόταση της Κομισιόν. Οι συνομοθέτες ήδη πέτυχαν πολύ πρόοδο. Το Κοινοβούλιο επί της αρχής τις τα πρόστιμα, την ευθυγράμμιση άλλε νομοθετικές πράξεις για τα φάρμακα, ενώ το Συμβούλιο ε, στήριξε κάποιες από τις τροπολογίες μας. Όμως υπάρχουν κάποια λεπτά ζητήματα που αφορούν τα έσοδα, το ταμείο, το αποθεματικό ταμείο διάλογο. Χθες, τώρα, πάντα πει, με την Βουλγαρική Παιδεία είχαμε τον πρώτο ανεπίσημο τριμερή διάλογο για τον κανονισμό για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Καλύψαμε τα βασικά της πρότασης ε, ε, και τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου, ακούσαμε την άποψη του Συμβουλίου, Κοινοβουλίου. Συζήτησε τώρα για τα πολιτικά πιο λεπτά ζητήματα, όπως είναι το thematic block για την καταπολέμηση μικροβής αντοχής, αποφάσεις για την άρνηση των διών κυκλοφορίας και συλλογή στοιχείων για τα αντιμικροβιακά φάρμακα χρησιμοποιούνται σε ζώα, τεχνικό επίπεδο. Τρίτος, ε, ο δεύτερο συγγνώμη τερμινή διάλογο προβλέπεται για τι 26 Φεβρουαρίου και η τεχνική συνάντηση θα προηγηθεί. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο τη Μερσιά διάταξη που είναι ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Διευθύντρια του ECDC για την όσο του ΛΑΙΜ. Και λοιπόν, λυπούμε στο συγγνώμη. Αυτή τη φορά θα ξεκινήσει ο κύριο Ράιμ, γενικό διευθυντή από τη ΓΑΜΑΔΕΛΤΑ ΣΑΝΤΕ. Ναι, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες εκτίθενται σήμερα στον κίνδυνο της ασθενείας ε, του Λάιμ. Η συναδελφός μου, η Δόκτωρα Μόν, ε, σύντομα θα κάνει μια παρουσίαση για την επιδημιολογία και τα νούμερα. Και οι δύο παρουσιάσεις μας προκρίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορούν όλα τα κράτη-μέλη ασθένεια του ΛΑΕΜ ανησυχεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια από τις πιο διαδεδομένες μολυσματικές ασθένειες στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Η γεωγραφική της κατανομή επίσης ε, μεταβάλλεται και γεωγραφικά πλάτη θα συμβάλλει σε αυξημένη διάδοση της ασθένειας σε ενδυμικές περιοχές. Παρότι λοιπόν δεν είναι νέα ασθένεια, η ασθένεια του ΛΑΕΜ Θεωρείται ότι μια ακριβή ε, περιγραφή τρόποι δεν μπορούν να συγκριθούν γιατί είναι διαφορετικά τα διαγνωστικά τεστ που χρησιμοποιούνται. Τρίτον, οπότε τα στατιστικά στοιχεία δεν βασίζονται σε τυποποιημένους ορισμούς. Επίσης δεν είναι τυποποιημένα τα συστήματα συλλογής δεδομένων. Παρ' όλα αυτά, η νόση αυτή αποτελεί παράγοντα σχέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην επόμενη διαφάνεια είναι η απόφαση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου 1082 του 2013 που δημιουργεί ένα δίκτυο κρατών μελών για την επιδημιολογική εποπτεία των νόσων. Ελέγχεται από, την, από το ECDC ώστε να δημιουργηθούν συγκρίσιμα και σύμφωνα που μας καθορίζουν ε, για ποιε ασθένειε θα συλλέγουμε δεδομένα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 51 τέτοιε ασθένειε υπό ευρωπαϊκή επιτήρηση. Και ο κατάλογο αυτό, και αυτό είναι το σημαντικό που θέλω να σα πω σήμερα το πρωί, ο κατάλογο των νόσων αναθεωρείται αυτή και εξετάζεται το κατά πόσο η νόσο Lyme θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις, ε, ε, στο μέλλον στις ε, μεταδοτικέ ασθένειε και ανάπτυξη εμβολίων. Τέλος, 25 εκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί στο πλαίσιο της Ευρω... πρωτοβουλίας ευρωπαϊκής ε, χρηματοδότησης για καινοτόμους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ειδικά για την ανάπτυξη ενός εμβολίου κατά της νοσουλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Άμον, παρακαλώ. Yes, thank you. Ε, ευχαριστώ. Εγώ θέλω να σας ε, δώσω λίγο πολύ κάποια ιστορικά, ιστορικές πληροφορίες, το υπόβαθρο όπως είπε και ο κύριος ε, από την Κομισιόν, πρόκειται για μία ε, λίμωξη βακτηριακή ε, που μεταφέρεται μέσω των τσιμπουργιών και δεν έχει να κάνει με την εγκεφαλίτιδα. Και πρώτο ανακαλύφθηκε το 77 από τον Λάιμ και μάλλον στο Λάιμ County στη ΣΥΠΑ. Και από εκεί πήρε και το όνομά του. Υπάρχουν διάφορα είδη βακτηρίων που δημιουργούν αυτή την νόσο λάιμα, αλλά μόνο ένα τσιμπούρι, ε, το εξόντες ρίξιμους, δημιουργεί προκαλευτίνος. Από πού μπορεί κανείς να κολλήσει. Από εκεί που έχει τσιμπούρια τους αρέσουν οι θάμνοι, το γρασίδι, θα τους βρείτε σε ανοιχτά βοσκοτόπια, σε θάμνους, σε δάση, όχι όμως μόνο στη φύση, αλλά και στα αστικά πάρκα ή στους κήπους, στα σπίτια σας. Δηλαδή η έκθεση είναι αρκετά μεγάλη, μπορεί κανείς να έχει. Η κλινική παρουσίαση, ε, τρεις ε, βασικά είναι φάση σε η πρόορη εμφάνιση, εκδήλωση που βλέπετε εδώ στην εικόνα αυτό το ερήθημα, ερήθημα migrants. Ε, είναι κόκκινο, έξω και όλο το ερήθημα και migrants γιατί ε, μεταφέρεται, μεταναστεύει στο ε, δέρμα και σε άλλες περιοχές. Δεν χρειάζεται κάποια εργαστηρική δοκιμή. Αντιβιωτικό αρκεί. Αλλά δεν είναι πάντοτε τόσο ξεκάθαρο, δεν υπάρχει πάντα αυτό το σύμπτωμα και οι διαγνωστικές δοκιμές δεν είναι τόσο ευαίσθητες και έτσι προκύπτει και το πρόβλημα. Γιατί πάει μετά στην επόμενη φάση που είτε έχουμε οξία νευρολογική, καρδιακή ε, συμπτωματολογία και έχουμε τελικά την ε, νόσο Lyme. Και υπάρχει και ένα τρίτο, είναι όψιμη εμφάνιση της νόσου, που θεωρείται η όπως μάλλον η επίμονη αρθρίτιδα. Η επιδημιολογία δεν είναι γνωστή ιδιαίτερα. Διότι τα στήματα επιτήρησης ε, μεταξύ των χώρων της Ένωσης ε, διαφέρουν. Και οι προσπάθειες που είπε και ο Τζον ε, που γίνονται ακριβώς στο στόχο αυτό έχουν την εναρμόνιση ε, έχουμε κάνει μια μεταανάλυση όλων των δεδομένων που είναι, είναι ήδη διαθέσιμα εδώ και 25 χρόνια. Υπάρχει και μια βιβλιογραφική επισκόπηση, 11,5 άνθρωποι ανά 100.000 προσβάλλονται. Αυτό είναι το στοιχείο. Βέβαια υπάρχει διακύμανση στη βιβλιογραφία ένας ή και 100 ανεκατό χιλιάδε. Δηλαδή υπάρχει μια ευρία γκάμα ε, διαφορετικών πληροφοριών. Χρειαζόμαστε στοιχεία στα οποία μπορούμε να βασιστούμε. Σε ό,τι αφορά τη διάγνωση, είναι ένα ιολογικό τεστ αυτό που γίνεται. Και εδώ έχουμε μια συστηματική επισκόπηση, είναι σαφές ότι η ευαισθησία στις πρόορες φάσεις είναι χαμηλή σε ό,τι αφορά ε, την ηλικία 5% περίπου σημαίνει ότι το 5% αυτών που έχουν προσβληθεί δεν ανοιχνεύονται σε αυτό το στάδιο. Και αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο λέμε ότι χρειάζεται καλύτερα διαγνωστικά τεστ. Όσο καλύτερη είναι η διάγνωση, μάλλον ε, η διάγνωση βελτιώνεται όσο η νόσος έχει προχωρήσει, αλλά και εδώ τη θεραπευτική αντιμετώπιση είναι πιο δύσκολη. Δεν υπάρχει εμβόλιο. Υπήρχε ένα που αποσύρθηκε το 2002, επειδή υπήρξαν διάφορες ανησυχίες παρότι δεν αποδείχθηκε ότι υπήρχε κάποια σχέση μεταξύ του εμβολίου και της ε, αρθρίτιδος ε, στην ε, μελέτες ασφάλειας φάσης 4. Έχουμε τώρα κάποια υποψήφια νέα εμβόλια, έχουμε δοκιμές φάσης 1 στη ΣΥΠΑ και στο Βέλγιο. Όταν λέμε φάση 1 σημαίνει ότι είναι η πρώτη φάση, άρα θα πάρει χρόνια και μίλησε για χρηματοδότημα από την Ένωση Project και ο Τζον. Τι μας απομένει λοιπόν η αποτροπή, δηλαδή να μην μας δαγκώσει τσιμπούρι ή αν μας έχει δαγκώσει να το αφαιρέσουμε ώστε το πιο γρήγορα αλλά με ασφάλεια από το δέρμα μας. Και γι' αυτό υπάρχουν και κάποια οδηγίες για το πώς μπορούμε να προστατευτούμε από τα τσιμπούρια και πώς να τα αφαιρέσουμε. Πρέπει να γίνει αυτό το συντομότερο δυνατό γιατί όσο πιο πολύ μένει στο δέρμα μας το τσιμπούρι τόσο περισσότερο αυξάνεται ε, η πιθανότητα να μεταδώσει αυτό το βακτήριο. Αν δεν είναι επιτυχής αυτή η αφαίρεση. Υπάρχει θεραπευτική αντιμετώπιση με τα αντιβιωτικά και το καλό νέο είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει να υπάρχει μικροβιακή αντοχή. Θα πρέπει να πάρει ε, με έγχυση τα αντιβιωτικά ο ασθενής. Το ίδιο και στην όψιμη Line. Από το 11 και μετά προσπαθήσαμε να καταλήξουμε σε κάποια συνένεση ό,τι αφορά την επίσης ε, δημοσιοποίηση κάποιες επιστημονικές συμβουλές για την επιδημιολογία και για την ε, χωρική επέκταση της νόσου Λάιμ και επισκοπούμε συστηματικό στη βιβλιογραφία σε ό,τι αφορά τη διάγνωση και τις εργαστηριακές δοκιμές. Και βλέπετε εδώ σε αυτή τη διαφάνεια όλα ακριβώς αυτά τα υλικά, τα έντυπα. Έχουμε βέβαια και αυτές τις, αυτά τα φυλάδια με κάποιες εικόνες και κάποια δυνατά για να βλέπουμε ε, την σχέση και τα, τις αντιστοιχίες ή αναντιστοιχίες της ε, λόγω νόσου σε σχέση με άλλες μεταφερόμενες από τη Συμπουργία Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσω το λόγο στα μέλη τώρα. Εάν θέλετε να μιλήσετε, πείτε. Ευχαριστώ και του εισηγητές για τι δύο παρουσιάσει του. Νομίζω ότι πολλοί χαίρονται που, θα, που έχουμε συμπεριλάβει το θέμα αυτό στην ημερήσια διαταξή μα στην Επιτροπή ότι δεν μπορώ παρά να πω ότι στην Ιρλανδία υπάρχει και η οργάνωση TikTok που προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει για το όλο θέμα και να καλλιεργήσει την οτροπία όσοι έχουν την όσο να ζητήσουν διάγνωση. Ε, ερώτηση λοιπόν και να τις θέσω τις ερωτήσεις μου εκ μέρους όσων ήρθαν σε επαφή μαζί μου. Έχουν ε, σε ευρωπαϊκά και αμερικανικά ε, εργαστήρια δεν γίνονται δεκτά. Ε, και επίσης για την ευαισθητοποίηση και την γνώση περί αν μπορούν να προτείνουν μια θεραπεία. Επίσης δεν γνωρίζουν καν να κάνουν τη σωστή διάγνωση. Επίσης για την κατάσταση της νόσου. Ακούω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χαίρομαι ότι θα αναθεωρηθεί ο κατάλογο και πολύ σύντομα θα υποβληθεί σχετική πρόταση. Διότι είναι πολλοί αυτοί που αυτή τη στιγμή υποφέρουν και κάποιοι δεν γνωρίζουν καν ότι έχουν. Του επαγγελματίε ή σε όσου ασχολούνται με τι δραστηριότητε ψυχαγωγία, όπου μπορεί κανεί να δεχθεί πιο εύκολα επίθεση από τσιμπούρια. Πρέπει λοιπόν να έχουμε τη σχετική ενημέρωση και ελπίζω με τι παρουσιάσει σα να κάνουμε κάποια. Ναι. Και τώρα η κυρία Κλούν. ξέρω που κάθεται, αλλά έχει και το λόγο. Κυρία Κλούν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι άκρος σημαντικό το θέμα. Στην Επιτροπή. να αντιβιωτικά, ναι ή όχι και για τις διάφορες μελέτες που χρηματοδοτούνται για τα διαγνωστικά στα εργαστήρια. Αυτό είναι πρόβλημα αυτή τη στιγμή, διότι οι δοκιμές που έχουμε αυτή τη στιγμή ε, έχουν να κάνουν μόνο με τα αντισώματα. Και το πρόβλημα είναι να εξαπλωθεί ακόμη περισσότερο, να δεγκωθεί ακόμη περισσότερο ο αριθμός των κρουσμάτων. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, πώς μπορούν αυτές οι νέες δοκιμές και αυτά τα τεστ να προχωρήσουν γρηγορότερα. Μήπως χρειαζόμαστε χρηματοδότηση και για τη διάγνωση και ταυτόχρονα για την διάγνωση σε και περισσότερες, περισσότερους πόρους για τη θεραπεία. Θέλουμε η βορελίωση να αντιμετωπιστεί. Θέλουμε να υπάρξει συνεργασία σε διεθνέ επίπεδο οι δυνατόν. Γιατροί από όλο τον κόσμο να ενώσουν τι δυνάμεις του και να δημιουργήσουν κοινέ ομάδε φορεί που να ασχοληθούν. Αυτό είναι ο σωστό δρόμος να δοθεί μεγαλύτερη ε, προσοχή στην Όσο ΛΑΙΜ. Για 20 χρόνια ε, διαγνωζόταν ε, η κατάσταση αυτή εγκαίρως και μάλιστα έχει οδηγήσει και σε ανάγκη μεταμόσχευσης καρδιάς. Τα πράγματα, το εμβόλιο για τα, κατά τα δείγματα εντόμων νομίζουν ότι είναι προστατευμένα, αλλά δεν ισχύει το ίδιο. Και και από όσου ε, διαχειρίζονται φυσικά πάρκα ε, έχουμε ακούσει και πρέπει να είναι έννοια και όλα αυτά τα οποία μας είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ένα βήμα γίνεται νομίζω σήμερα για να μπορούμε να ενημερωθούμε καλύτερα, να λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα για να μπορέσουμε να μειώσουμε την επίπτωση της νόσου λάιμ. Ευχαριστώ κύριο Σπότς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε ξέρουμε πώς να προστατευτούμε και πώς να το αντιμετωπίσουμε. Uh, uh, Από παραστολόγους, uh, γιατρούς και άλλους συναδέλφους περιοχές που δεν ήταν μέχρι τώρα παρούσα. Και βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει ευαισθητοποίηση, αλλά πρέπει το φορέα να παρακολουθούμε. Πού πάει. Thank you πρώτες ε, φάσεις ε, έγινε διάγνωση νόσου του Λάιμ και μετά ε, άλλαξε η διάγνωση σε κάτι άλλο το οποίο δεν μπορούσε να θεραπευτεί. Νόσο του παρακαλώ. Έχετε το λόγο κύριε Ράν. Η συζήτηση αυτή δείχνει ότι υπάρχουν πολλές ε, συνδέσεις μεταξύ της νόσου του ΛΑΕ. Είναι διάφοροι οι παράγοντες ε, και αυτό που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε εδώ είναι το να τυχές αυτού του ζητήματος της ε, νόσου του ΛΑΕΜ είναι ότι μεταφέρεται από φορέα και ότι μεταβάλλεται με το χρόνο. Και μιλήσαμε για τα ποσά, μιλήσαμε για 40 εκατομμύρια ευρώ για την έρευνα, οπότε έχουμε αυξημένη στη σωστή κατεύθυνση, αλλά το πρώτο πρέπει να κάνουμε θα είναι να καθιερώσουμε ένα καλό ένα σύστημα επιτήρησης και αυτό θα οδηγήσει και του εθνικό επίπεδο να αναζητήσει περαιτέρω